Som Καλώς ορίσατε στη συνεδρίασή μας. På punkten 1. Eh- Αρχίζουμε αμέσως στην ημερήσια διάταξη και πάμε στο πρώτο σημείο αυτή. Πρόκειται για την έγκριση τη ημερήσιας διάταξη φυσικά. Δεν έχουμε εδώ κάποιε προτάσει, ενστάσεις και επομένως εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Κατευθείαν το σημείο 2, η πρώτη συγκοινώση του Προέδρου. Πρώτα-πρώτα, έχω να σα πω το εξή. από την 1η Μαΐου θα έχουμε καινούργια προσταμένη της ε, γραμματείας, καλώς όρισα. Έχουμε στο παρελθόν συνεργαστεί πάρα πολύ αρμονικά και επομένως καλώς όρισε στην γραμματεία μας. Επίσης, τον Εμίλ Ντουάρ να ευχαριστήσω ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα του τμήματάρχη μέχρι σήμερα και με εκείνον ήταν πάρα πολύ θετική η εμπειρία της εργασίας. Πρώτη για μια μεταβατική περίοδο που πήγε πάρα πολύ καλά και επομένω από τη νέα του θέση στη γραμματεία πάλι με χαρά θα συνεργαζόμαστε. Το επόμενο. Όταν αποφασίσαμε να καταρτήσουμε αυτή τη μέση διάταξη, θεωρήσαμε ότι δεν έχουν πάρα πολύ χρόνο στην ε, ε, διάθεσή μας, οπότε είπαμε η κυρία Μποσκούρτ να, να πει αύριο τα δικά της, το, το δικό της σημείο να το αναπτύξει, οπότε ε, αυτό και θα γίνει, θα συζητήσουμε το σημείο της κυρίας Μποσκούρτ αύριο. Τώρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό να οργανίσει συνεδρίαση, σημαντικό για όλους τους βουλευτές. Δηλαδή αύριο στις 9 θα αρχίσει η συνεδρίαση και όχι στι 9 και 10, όχι στι 9 και 7, ούτε στις 9 και 4, ούτε στι 9 και 2. Θα ξεκινήσουμε στις 9 ακριβώς. Τώρα, στις 9 το παράδειγμα θα αρχίσει και όποιο δεν είναι εδώ, κακό του κεφαλιού του. Δεν θα σας πω τίποτα άλλο, γιατί θα πρέπει να διεξέλθουμε ένα σωρό θέματα και θα πρέπει να ψηφίσουμε ένα σωρό θέματα, οπότε και αυτό θα γίνει. Θα αρχίσουμε ακριβώς στις 9. Ξέρετε ότι είμαι Σκανδιναβός και επομένω ξέρετε ότι είμαι συνεπής σε όλα αυτά. Δεν θα περιμένω κανένα για να ξεκινήσω. Το επόμενο σημείο τώρα είναι το σημείο παριθμών 3. Τα πρακτικά της συνεδρίασης των συντονιστών της 27 Μαρτίου. Αν δεν έχετε καμία αντίρρηση, τότε σας προτείνω να εγκρίνουμε τα πρακτικά αυτής της συνεδρίας των συντονιστών. Σύμφωνοι, οπότε πάμε τώρα στο πρώτο ουσιαστικό πολιτικό σημείο. Θα γίνει ανταλλαγή απόψεων με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διασώτα των φίλων. πρώτα πρώτα δώσουμε τον ε, οργανισμό στην προσταμένη του Οργανισμού Θεμελιών Δικαιωμάτων και κατόπιν τις τελούσεις ε, καθήκοντα διευθυντού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πάρα πολύ την ε, Επιτροπή Δημάτων Γυναικών και Ισότητας των Φίλων που μας δίνει σήμερα την ευκαιρία να σας τα πούμε. Θα είμαι όσο σύντομη μπορώ. Και κατόπιν η συνάδελφο θα συνεχίσει. Οπότε, πρώτα-πρώτα, για τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σε σχέση με την βία κατά των γυναικών και τη σχετική έρευνα. Με λίγα λόγια, πρώτα-πρώτα, ζητήθηκε να γίνει αυτή η έρευνα το 2009 υπό Ισπανική Προεδρία. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ισότητας και βέβαια τον Νοέμβριο του 2009 ε, είχαμε το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, το οποίο είχε ζητήσει επίση να συλλέξουν αυτά τα δεδομένα. Αυτό είναι επομένω το ιστορικό πλαίσιο για το έργο που επιτελέσαμε. Και με λίγα λόγια, η δουλειά μα είναι έρευνα. Έρευνα για ε, το, το, το, το χώρο, για, για το χώρο δουλειάς και <clears throat> για την ε, έρευνα έξω στην κοινωνία, εκεί όπου έχουμε ένα κενό στα δεδομένα που έχουμε, σε σχέση με τα δεδομένα που έχουν τα αρμόδια υπουργεία και η ποινική δικαιοσύνη και ξέρουμε όμως από παλαιότερες έρευνες, όπως και εσείς ξέρετε, ότι τα έρευνα, η έρευνα, τα στοιχεία για την βία των γυναικών, αυτά τα στοιχεία πάσχουν σε αρδιότητα, για την πέμπτη έρευνα που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα στον Οργανισμό Θεμελιδών Δικαιωμάτων. Επομένω, πρόκειται για μία μόνο τη έρευνα που έχουμε κάνει και η άλλη αφορούσε τι λεσβείε και ομοφιλόφιλους ε, σε σχέση με τη δυσμενή διακρίση τη βάρο των προσώπων. Ακόμη. Σε ενωσιακό επίπεδο δεν έχουμε κάποια έρευνα που να καλύπτει αυτό το οποίο θέλουμε, οπότε και εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο και τους όμως επόμενους μήνες πρόκειται να δοθεί στη δημοσιότητα. Βεβαίω και πρόκειται για ένα τομέα όπου έχουμε καταπάτηση των θεμελιωτών δικαιωμάτων. Για να τι έχουμε που έχει φτάσει η κατάσταση, οπότε όταν ρίχνουμε μια ματιά στις υπάρχουσες έρευνες, διαπιστώνουμε ότι αυτές για τη βία κατά των γυναικών, όπως γνωρίζετε, καλύπτουν πάρα πολύ μικρό βαθμό συγκρισιμότητας. Το Συμβούλιο της Ευρώπης επίσης είχε ξεκινήσει μια τέτοια έρευνα, το ΟΗΕ και επομένως ε, και σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν τέτοιες έρευνες, αλλά δεν υπάρχει συγκρισιμότητα μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης, γιατί διαφέρει η νομοθεσία, ο η μέθοδος συλλογής ε, δεδομένων, και, και όταν επομένω έχουμε το συμπίλημα των δεδομένων δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε. Και, εάν θυμάμαι καλά, καλύπτουμε τέσσερα κράτη-μέλη. Μόνο. Οπότε μόνο αυτά τα τέσσερα κράτη-μέλη μπορούν να συγκριθούν. Όμως, έχουμε διάφορες άλλες ε, ε, όπως του, του, του Συμβουλίου ΕΠΣΚΟ που, αφορούσε την ε, κρίζωση της βίας και των ηλιακών δεν υπάρχει εδώ συγκρισμότητα επομένως. Επομένως, έχουμε κάποιους δείκτες του Συμβουλίου της Ευρώπης, ε, κάποιες μελέτες του ΟΗΕ και οπότε εμείς προσθέσουμε όλα αυτά να τα συνδυάσουμε και του πάτου προσώπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έγινε. Προσπαθήσαμε να δούμε τότε κάθε τέτοια έρευνα θα πρέπει να είναι χρήσιμη για να χαράξουν πολιτική. Θα πρέπει να βρουν κάποια στατιστικά τα οποία να χρησιμοποιούνται σαν ε, δείκτες, κριτήρια. Οπότε έτσι να λέμε ότι έχουμε συγκρίσιμα δεδομένα τα οποία μα δίνουν αυτού του δείκτε και ο κόσμο μπορεί να διαπιστώσει σε ποιο σημείο βρίσκεται η κατάσταση σε κάθε κράτο μέλο ή σε κάθε κράτο μέλο σε σχέση με άλλο κράτο μέλο ή τρίτο κράτο. Βεβαίω και έχουμε την ΕΠΣ, του, του Συμβουλίου ΕΠΣΚΟ και έχουμε και κάποιες ε, άλλες ε, ε, και και αιτήματα από μέλη και θα σας πει που αλλού χρειάζονται αυτά τα δεδομένα και οι συνάδελφος. Τώρα για να δούμε το κυρίως το κύριο τμήμα της έρευνας λέμε ότι οι βασικοί στόχοι της έρευνας είναι να προκύψουν αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα όσον αφορά την διάρκεια των γυναικών. Και για πρώτη φορά καλύπτουμε το σύνολο της Ένωσης. Ο Οργανισμός των Δικαιωμάτων ε, και κάνει αυτή την έρευνα κατόπιν ε, συνένεση που μορφώθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο μας πήρε κάποιο χρόνο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε αυτό το στάδιο της ολοκλήρωσης της μελέτης, γιατί πρόκειται περί αρκετά περίπλοκου εγχειρήματο. Άρα είπαμε ότι πρέπει να είναι χρήσιμα αυτά που βγάζουμε για τη της πολιτική, ούτω ώστε να έχουν πολιτικέ και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Επομένω, είπαμε ότι σε μελέτε μεγάλη κλίμακα έχουμε μεγάλη πείρα και δεν λέμε τώρα τον, στον ερωτηματολόγιο μα, αλλά είπαμε να βγαίνουμε στον δρόμο για να μιλάμε στις γυναίκες για την εμπειρία του σχετικά. Είχαμε δείγμα πάνω από 20.000 προσώπων σε άλλε μελέτε μας. Και τώρα, επομένω, κάτι τέτοιο κάνουμε όσον αφορά τη βία των γυναικών. Το χρονοδιάγραμμα ξεκίνησε το 2009 το πρώτο αίτημα και κάναμε επομένω αυτή τη ε, δοκιμαστική μελέτη το 2011. Δηλαδή ήθελα να κάνουμε και κάποιες γνωστικές συνεντεύξεις με, σε εστιασμένες ομάδες για κάποιους οι οποίοι είχαν πέσει θύματα βίας σε σχέση με βασικές έννοιες της έρευνας και επίσης ξεκίνησε η καθεαυτού έρευνα και η συλλογή δεδομένων το 2012, όπως είπαμε σε όλα τα κρατημέλη και την Κροατία. Ιδέα ανάλυση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων θα γίνει το 2013. Αυτά για το χρονοδιάγραμμα της έρευνας. Οπότε, με λίγα λόγια, έχουμε 27 κράτη-μέλη και την Κροατία. Συνολικά έχουμε 40.000 γυναίκες ε, με τις οποίες συνομιλούμε στα 27 μέλη και στην Τώρα τώρα μπορεί να μπορεί να το, το πώ είναι σχεδιασμένη, δομημένη η έρευνα. Τυχαία δείγματα, τυχαίο δειγματισμό γυναικών, αυτό είναι η έρευνά μα. Δεν πάμε σε κυβερνήσει οργανώσει, ούτε πηγαίνουμε σε φορεί εκεί όπου οι γυναίκε καταγγέλουν τη βία. Πάμε σε τυχαία πρόσωπα εκείνοι να μας πούν επομένω τι εμπειρία έχουν από πλευρά βία. Μιλούμε σε γυναίκες που είναι 18 ή πιο μεγάλες. Επίσης, ε, τα δεδομένα κατά ηλικία, παιδεία, απασχόληση, εθνική προέλευση, το αν ε, προέρχεται κάποιος ε, από άλλη χώρα, για μετανάστε κλπ. Ένα πρόσωπο ανά νοικοκυριό. Όλες οι συνεντεύξεις γίνονται πρόσωπο με πρόσωπο, ζωντανά ας το πούμε, και η διάρκεια είναι κατά μέσο όρο 50 λεπτά. Πολλές από αυτές είναι συντομότερες. Δεν έχει κάποια γυναίκα να αναφέρει αρκετά και άλλο έχουν φτάσει σε 2,5 Ωραία, στη συνέντευξη, εκεί που είχε πολλά να πει κάποια κοπέλα, κάποια γυναίκα. Είναι τυποποιημένο το ερωτηματολόγιο και επίσης έχει γίνει ακριβής μετάφραση, ούτως ώστε να χρησιμοποιήσει όλα τα μέλη. και τις συνέντευξεις τις παίρνουν κάποιες γυναίκες, κοπέλες, οι οποίε έχουν εξειδικευμένη κατάρτιση και εκπαίδευση. Περιεχόμενο. Μόνο, μόνο γενικά θα ήθελα να σας πω καλύπτει την ε, σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βία. Επίσης καλύπτει νέες ή πρόσφατα ανεγνωρισμένες μορφές βίας, ε, ας πούμε νέες μορφές είναι το να στέλνει κανείς, να κανείς βία στέλνοντας email ή μηνύμα στο κινητό τηλέφωνο. Επίσης εξετάζουμε την ε, βία από τους συντρόφους αλλά και από τρίτα πρόσωπα. Επομένω, τα πρόσωπα με τα οποία έχει κάποια γυναίκα κάποια σχέση, αλλά και όχι. Επίσης, στο, στο χώρο εργασίας, στο σπίτι και αλλού. Εκεί να δούμε ποιος έφταγε. Λοιπόν, σε όλους αυτούς τους χώρους, επίσης, τους ζωτούμε να μας, τις μας πούνε το εάν ξέρουν τα δικαιώματά τους για να γνωρίζουν τι υπηρεσίες παράσχονται, για να τις βοηθήσουν επίσης για το πώς τις καθιστούν θύματα στην ε, παιδική ηλικία. Βάσει των αναμνήσεών τους, διότι ο οργανισμός των δικαιωμάτων ε, ασχολείται και με τους ανηλίκους. Οπότε καλύπτονται, καλύπτονται και τα δεδομένα που αφορούν την παιδική ηλικία των γυναικών. Επίσης, την υπόλοιπη ζωή και τι έγινε τους τελευταίους 12 μήνες σε σχέση με το τι πολιτικές σα Επίσης, για το κατά πόσον καθυποτροπή υποτροπή έχουν υποστεί αυτού του είδους την, τη βία, κατά πόσο έχουν γίνει θύματα, κατά επανάληψη. Παράδειγμα επίσης των όσων συζητούμε είναι οι συνέπειες της βίας, αυτές δηλαδή που έχουν υποστεί βία, ρωτούμε τι τραυματισμό έχουν υποστεί, εάν έπρεπε να σταματήσουν να δουλεύουν, εάν ήταν ε, παρόντες και ανήλικοι, όπως όταν έγινε από τον σύντροφό τους κλπ. Επίσης ρωτούμε, με ποιον ήρθαν σε επαφή μετά, με την αστυνομία Φερρυπίν, αν είναι ικανοποιημένες από τη βοήθεια που τους παρήχθη. Επίσης, εάν δεν κατήγγυλαν την άσκηση βίας, για ποιους λόγους δεν ήταν σε επαφή με κάποιες υπηρεσίες, με κάποιες, ας πούμε την αστυνομία, οπότε βλέπουμε εδώ πέρα τα, τα, τα άδειλα στοιχεία, αυτά που δεν μας για την άσκηση της βίας. Επίσης, ποιος βοήθησε με κυβερνικές οργανώσεις μέσα σε ένα κράτος μέλος. Αυτά με λίγα λόγια ήθελα να σας πω, όμως τώρα θα πρέπει να σας, να σας ε, συμπληρώσω το ότι πάρα πολύ βοήθησε την έρευνα. Τα όσα είπαν οι εμπλεκόμενοι, οι Άγγοι, ας πούμε, το Ευρωπαϊκό του για των Φίλων, μας βοήθησε πολύ και, και άλλοι εμπειρογνώμονες από αλλού, όπως η Σίλβια, και εκτιμήθηκε πάρα πολύ η βοήθειά τους. Κάτι άλλο πρέπει να διευκρινίσω. Η έρευνα δεν μπορεί να τα καλύψει όλα. Σε μια έρευνα του γενικού πληθυσμού των γυναικών δεν μπορούμε να καλύψουμε κάποιες συγκεκριμένες μορφές βίας όπως τον σεξουαλικό γενετήσιο ακροτηριασμό διότι αυτό αφορά συγκεκριμένα πρόσωπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση άρα χρειάζεται μια πολύ στοχευμένη έρευνα για να το ψάξει αυτό προτυπώμες για πολύ συγκεκριμένες μορφές βίας κατά συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού δεν είναι δυνατόν μόνο σε γενική έρευνα όλα αυτά να τα καλύψει. Αυτό που το οποίο κάναμε ήταν. Θέλουμε να δούμε τι γενικότερε τάσει. Δεδομένα, το οποίο μπορεί να προκύψουν με διάφορου τρόπου εδώ που θέλουμε και κάτι άλλο, είναι και κάποια άλλη εκθέση που να κάνουμε που αφορά το κόστο της βίας κατά των γυναικών, ας πούμε, το κόστος που το οποίο πρέπει να φέρει η κοινωνία με το που δεν αντιμετωπίζει τη βία των γυναικών από πλευράς θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά και από πλευράς των ε, ημερών που, θα, δεν μπορούν να δουλέψουν οι γυναίκες, πρέπει να νοσηλευθούν κλπ. κλπ. Να, επομένως, πώς μπορούμε επίσης να βρούμε τα αποτελέσματα. Και σας ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κούντι. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Ρέγκερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και σας και την Επιτροπή που δίνετε το λόγο στο Ινστιτούτο για την Ισοτοδία Φίλων να τοποθετηθεί εδώ. Και ευχαριστώ και την εκπρόσωπο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για την παρουσίαση. Εγώ θα σας πω κάποια πράγματα που συμπληρώνουν ε, τη δουλειά του οργανισμού. Εγώ θέλω να επικεντρωθώ στο χρόνο που έχω σε πολλές άλλες έρευνες ε, που το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων ε, υλοποιεί σε σχέση με την βία λογοφύλου. Εδώ βλέπετε αυτή τη διαφάνεια, βλέπετε ένα κατάλογο και θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ σε κάθε ένα στοιχείο. Καταρχήν, το πρώτο σημείο αφορά τις έρευνες για την υποστήριξη των θυμάτων στο πλαίσιο της ε, παρακολούθησης της ε, εφαρμογής της πλατφόρμας ε, για δράση στις χώρες που ανήκουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ξέρω ότι πρόσφατα λάβατε την έκθεση του ΑΕΚΕ που αναπτύχθηκε για την Προεδρία της Δανίας για την κλιματική αλλαγή. Η προηγούμενη έκθεση μας αφορούσε τη συμφιλίωση μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματική ζωής που έγινε για την Πολωνική Προεδρία. Τώρα αρχίζουμε να εργαζόμαστε και να υποστηρίζουμε την Προεδρία της Κύπρου γιατί αποφάσισαν να παρακολουθούν ε, την εφαρμογή ε, της ε, πλατφόρμας σε ό,τι αφορά την υποστήριξη των θυμάτων. Όπως ξέρετε, το 2002 η Προεδρία της Δανίας έδωσε κάποιες συστάσεις για 13 δείκτες στον τομέα της προστασίας των θυμάτων και εκεί καλυπτόνταν διάφορες υπηρεσίες σε αυτό το τομέα και αυτό που κάνει το Ινστιτούτο αυτή τη στιγμή είναι να παρακολουθεί την πρόοδρο στον τομέα αυτών των υπηρεσιών για τα θύματα της οικογενειακής βίας ε, κατά βίας κατά των γυναικών. Άλλη μια έρευνα η οποία ε, ουσιαστικά επεκτείνει την υποστήριξή μας ε, στην Προεδρία σε ό,τι αφορά τη συλλογή βελτιστών πρακτικών στην υποστήριξη των θυμάτων είναι ε, μία βάση δεδομένων για τις πηγές για την ε, σεξουαλική βία και μία ευρύτερη έρευνα για τι ε, τον ακροτηριασμό των γενετικών οργανών στις γυναίκες προσπαθεί να συλλέξει δεδομένα στα 27 κράτη-μέλη και στην Κροατία και επίσης έχουμε και μία έρευνα για τη συλλογή διοικητικών γενομένων για το GBV και συμπληρώνει την έρευνα που υποστηρίχθηκε προλίγου, που παρουσιάστηκε προλίγου. Το κύριο αντικείμενο της μελέτης, ε, όπως σας ανέφερα, ε, για την Κυπριακή Παιδεία είναι να υποστηρίξουμε τις υπηρεσίες για τις γυναίκες που είναι θύματα οικογενειακής βίας. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας τι θα κάνουμε, θα αναθεωρήσουμε τις ε, διάφορες έρευνες στην Ευρώπη σχετικά με τα ποσοστά της επικράτησης, αλλά όπως αναφέρθηκε ήδη, αυτές οι έρευνες, αυτές οι μελέτες έχουν ε, όρια σε σχέση με τη συγκρισιμότητα αλλά θέλουμε να δείξουμε τι έχει ήδη γίνει. Και επίσης ε, θέλουμε να δείξουμε ποια είναι τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το κράτος ε, στα 27 κράτη-μέλη και στην Κροατία για την εξάλληψη της βίας. Ένα δεύτερο σημείο που βλέπετε εδώ σκοπεύουμε εδώ στην συλλογή πρωτογενών ε, δεδομένων ε, σε ό,τι αφορά το βαθμό, τον αριθμό και την πραγματική χρήση ε, αυτών των υπηρεσιών υποστήριξης. Εμείς θέλουμε να αντικατοπτρίσουμε και την τυπολογία των υποδικτών που προτέθηκε από το Συμβούλιο το 2002 αλλάζει η πραγματικότητα και οι ανάγκες υποστήριξης αλλάζουν και υπάρχουν τώρα διαθέσιμες νέες υπηρεσίες, ε, υπηρεσίες που εγκρίθηκαν ε, το 2002 πριν 10 έτη, δεν είναι τόσο σχετικές σήμερα όπως ήταν πριν 10 έτη. Έτσι λοιπόν θα θέλαμε να ασκήσουμε μια κριτική σε αυτό το θέμα και να δώσουμε μια σαφή εικόνα των σημερινών αναγκών των γυναικών που είναι θύματα βίας. Ε, ένα άλλο σημαντικό σημείο που εστιάζουμε στη μελέτη και που θα το αντικατοπτρίσουμε εδώ όχι μόνο από ποσοτική αλλά και από ποιοτική σκοπιά είναι ο συντονισμός της, ε, των δημόσιων συστημάτων υποστήριξης ε, των θυμάτων οικογενειακής βίας και ακολουθώντας ε, τη βέλτιστη πρακτική, τις βέλτιστες που είχαμε σε προηγούμενες έρευνε, θέλουμε να ευστήσουμε την προσοχή των κρατών μελών, όχι μόνο στο ίδιο το θέμα, αλλά και στην ποιότητα των δεδομένων, ε, δηλαδή στα κενά των δεδομένων και να ε, χορηγήσουμε συστάσεις για τη βελτίωση της συλλογή των δεδομένων για την υποστήριξη των θυμάτων. Ένα άλλο σημείο εστίασης θα είναι η συλλογή εργαλείων, μεθόδων και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα αυτό. Μετά από διαβουλεύσεις εις βάθος με τα ενδιαφερόμενα μέρη καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αυτές οι εκθέσεις των προεδριών θα μπορούσαν να είναι πιο χρήσιμες και θα μπορούσαν ε, ε, να είναι πιο ε, αποτελεσματικές αν μπορούσαμε να επικεντρωθούμε στο τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη. Έτσι λοιπόν, αυτή η ευρύτερη προσέγγιση ε, σε αυτόν τον ε, τομέα της Προεδρίας όπως αποκαλείται θα εφαρμοστεί τώρα και η έκθεση αυτή θα είναι η πρώτη η οποία θα, θα, είναι η πρώτη η οποία θα περιλαμβάνει αυτή την ευρύτερη προσέγγιση επί του θέματος. Τώρα θα ήθελα να επικεντρωθώ στη μελέτη που έχει διολοκληρωθεί, στην έρευνα που έχει διολοκληρωθεί. Αλλά τώρα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα. Δεν επρόκειτο για μια μεγάλη μελέτη ως προς το παιδί εφαρμογή. Αφορούσε τη συλλογή δεδομένων ε, σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών. Ε, αλλά βάσει των δεδομένων που είχαμε στο Ινστιτούτο, αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε σε αυτό το είδος της βίας, ε, γιατί έχει μια κρυφή φύση και είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Λείπουν σε αυτό το τομέα τα δεδομένα η ιδέα της μελέτης ήταν να αναθεωρήσουμε τις πηγές των δεδομένων ε, στον τομέα της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών, να χαρτογραφήσουμε τους διάφορους πρωταγωνιστές και να οικοδομήσουμε μια βάση δεδομένων ε, δημόσιας πρόσβασης για όλα τα κράτη-μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το πεδίο της μελέτης εδώ το βλέπετε, βλέπετε πώς ορίστηκε σεξουαλική βία. Εδώ θέλω να αναγνωρίσω τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών. Βλέπετε εδώ ότι καλύψαμε την ε, σεξουαλική βία. Από τη μελέτη και τα αποτελέσματα θα τοποθετηθούν στη βάση δεδομένων και θα είναι διαθέσιμα για δημόσια πρόσβαση πάρα πολύ σύντομα, μέσω της ιστοσελίδας. Όπως ανέφερα, η βάση δεδομένων θα δώσει τη δυνατότητα να δούμε ε, ποια άλλα όργανα εμπλέκονται σε αυτό το τομέα, ποια είναι η βιβλιογραφία, ποιε είναι οι μέθοδοι που έχουν χρησιμοποιηθεί όταν εργαζόμαστε με τα θύματα. Και συγγνώμη που όλα αυτά τα αναφέρω τόσο γρήγορα. Τώρα, το θέμα του ακροτηριασμού των γεννητικών οργάνων των γυναικών. Όπως ε, ανέφερα, αρχίσαμε να κάνουμε αυτή την έρευνα βάσει αιτήματο της Κομισιόν, της Επιτρόπου Ρέντινγκ. Ο κύριος στόχος της έρευνας, της μελέτης, είναι να υποστηρίξουμε και να συνεισφέρουμε στην μελλοντική ανάπτυξη στρατηγικών για την καταπολέμηση διάφορων μορφών βίας κατά των γυναικών μέσω της ε, συλλογής δεδομένων για το θέμα του ακροτηριασμού των γεννητικών οργάνων στα 27 κρατημέλη και στην κρατία. Βλέπετε εδώ ότι θα χαρτογραφήσουμε τις εφιστάμενες πληροφορίες και δεδομένα σε ό,τι αφορά και τις πολιτικές σε το νομικό πλαίσιο, τους πρωταγωνιστές, τις μεθόδους και τα εργαλεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κροατία θα προβούμε σε μία εισβάθος ποιοτική ανάλυση των πρακτικών αυτών και των αιτιών τους και των πιθανών μελλοντικών τάσεων. Και επίσης θα εντοπίσουμε τα κενά ε, σε ό,τι αφορά τη συλλογή δεδομένων και θα δώσουμε συστάσεις για το πώς θα βελτιωθεί η συλλογή δεδομένων στον τομέα αυτό. Και τέλος, έχουμε μία νέα πρωτοβουλία η οποία συμπληρώνει πάρα πολύ καλά τη μελέτη που παρουσιάστηκε από την προλελήσασα. Πρόκειται για μια μελέτη που επικεντρώνεται περισσότερο σε διοικητικά δεδομένα, δηλαδή μιλάμε για διαφορετικές πηγές πληροφοριών για τη βία και το λόγο του φύλου. Και εδώ θέλουμε να θεωρήσουμε τα είδη και τις μεθόδους της συλλογής διοικητικών δεδομένων. Όπως βλέπουμε, τα διοικητικά δεδομένα δεν μας δίνουν μια πλήρη εικόνα ε, αυτού του είδους της βίας για διάφορους λόγους. Οι γυναίκες δεν είναι πρόθυμες ε, να καταγγείλουν τα περιστατικά και οι οργανισμοί που συλλέγουν αυτά τα δεδομένα, όπως πούμε το η αστυνομία ή τα δικαστικά συστήματα, δεν συλλέγουν τα δεδομένα με συγχρονισμένο τρόπο και υπάρχουν και άλλα προβλήματα που σχετίζονται με τα διοικητικά δεδομένα. Δεν αντικατοπτρίζουν πλήρω το μέγεθο του προβλήματο. Και θέλουμε λοιπόν να επιστήσουμε την προσοχή στο πρόβλημα αυτό. Επίση, σχεδιάζουμε να αξιολογήσουμε το εφικτό τη συλλογή συγκριτικών δεδομένων σε αυτόν τον τομέα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και το στατιστικό δυναμικό αυτών των πηγών. Τέλος, η βία κατά των γυναικών λόγω του φίλου τους θα είναι ένα σημαντικό τμήμα ενός σημαντικού καθήκοντος που είναι η οικοδόμηση του δίκτυ ισότητας των δύο φύλων. Εδώ έχουμε αναφέρει τους κύριους και η βία θα είναι ένας από τους ε, τομείς. Εδώ βλέπετε απλώς μία πρόταση. Θεωρήστε τη λοιπόν ως πρόταση εξακολουθεί να είναι υποεκπώνηση. Εδώ βλέπετε το κύριο πλαίσιο του δίκτυ και όπως βλέπετε η βία είναι ένα τμήμα. Λόγω περιορισμών που μας θέτουν τα στοιχεία, λόγω πολύ λίγων πηγών δεδομένων στοιχείων για την οικογενειακή βία, η βία δεν θεωρηθεί ως τομέας με τον ίδιο τρόπο όπως άλλοι τομείς. Εμείς είχαμε σκεφτεί εδώ, σκεφτόμαστε μάλλον διάφορες δυνατότητες για το πώς να το αντιμετωπίσουμε και η βία είναι και ένα πρόβλημα διαφορετικής φύσης κατά κάποιο τρόπο από το θέμα του πώς συμμετέχουν γυναίκες και άνδρες ε, στη λήψη αποφάσεων, ε, στην εργασία. Είναι ένα διαφορετικό πρόβλημα και γι' αυτό συζητάμε αυτή τη στιγμή τι θα κάνουμε αλλά ο στόχος μας είναι τουλάχιστον να το αντικατοπτρίσουμε ως ένα σημαντικό τμήμα της ισότητας των δύο φύλων και στο μέλλον όταν θα καλύπτεται από τα δεδομένα όπως ελπίζουμε θα είναι πάρα πολύ σημαντικό στομέα του δίκτυ όπως και οι υπόλοιποι τομείς. Αυτή είναι η σύντομη παρουσίασή μου και αν έχετε ερωτήσεις ευχαριστώ να σας απαντήσω. Σας ευχαριστώ. Eh, σας ευχαριστώ. Και τις ε, δύο μιλητές για τις παρουσιάσεις σας, ενδιαφέρουσες. Και θα ήθελα τώρα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση στο σημείο αυτό. Παρακαλώ. Κυρία Τσέσκοβα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα για την ευκαιρία που μας προσφέρετε και ότι έφτασα με καθυστέρηση και ζητώ συγγνώμη. Θα ήθελα να πω ότι ταυτόχρονα λαμβάνουν χώρα δύο διαφορετικές συνεδριάσεις επιτροπών και γι' αυτό χρειάστηκε να ε, ε, καθυστερήσω. Το θέμα το οποίο συζητούμε σήμερα με έχει απασχολήσει και στην Τσεχία, στην πατρίδα μου. Είχα την ευκαιρία μάλιστα ένα κομμάτι της παρουσίασής σας να το παρακολουθήσω μέσω του διαδικτύου. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Ε, το θέμα της οικιακής ή ενδοοικογενειακής βίας με απασχολεί ιδιαίτερος. Είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να αντιδράσουμε, θα πρέπει να αναλάβουμε δράση, θα πρέπει συνεχώς να το θίγουμε και να το συζητούμε και να το αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά. Αν και πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οτιδήποτε μέτρο και να εισαχθεί μόνο σταδιακό μπορεί να είναι, μόνο αργά-αργά μπορεί να φέρει καρπούς. Τώρα μια ερώτηση στη σχέση με τις ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις ε, που έχουν πολλές φορές συνεργασία και τα κράτη-μέλη. Υπάρχει λοιπόν αυτή η συνεργασία Ε, και στο, στο φθινόπωρο πέρυσι είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω σε μια σχετική εκδήλωση ε, από πρωτοβουλία της Τσεχικής Δημοκρατίας έγινε ένα μεγάλο συνέδριο όπου ε, ήρθαν διάφορες οργανώσεις για να συζητήσουν τα θέματα αυτά. Ήταν μάλιστα μεταξύ τους οργανώσεις οι οποίες προσφέρουν και άσυλο, ασφαλές καταφύγιο σε γυναίκες και κυρίως μητέρες με νεαρά παιδιά που πέφτουν θύματα αυτής της ενδοοικογενειακής βίας. Από την εκδήλωση αυτή είδα, όπως άλλωστε και πάλι στις εκδηλώσει, ότι οι οργανώσεις δεν έχουν αρκετά χρήματα στη θέση τους, δεν έχουν αρκετούς πόρους. όπως πολύ συχνά συμβαίνει. Και επίσης ότι τα καταφύγια αυτά δεν είναι πάντοτε επακριβώς προσδιορισμένα ως χώρο στον οποίο μπορεί να έχει καταφυγεί μόνο το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας. Δεν είναι αποκλειστική δηλαδή η διαμονή, αποκλειστικά ε, εξασφαλισμένη διαμονή για μια γυναίκα με τα παιδιά της ενδεχομένως που προσπαθεί να ξεφύγει από τον θήτη. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μεγάλες ανάγκες, ανάγκες σε βοήθεια ουσιαστική, αλλά και σε ε, βοήθεια τυπική. Και πρέπει να εξασφαλίσουμε συνθήκες ασφάλειας για τις γυναίκες με τα παιδιά τους, για όποιον πάει να, για όποιαν μητέρα καταφύγει εκεί, ώστε να μην έχει δικαίωμα ούτε καν να την επισκεφθεί ο σύζυγος Παύλα Θήτης, ε, όπως συμβαίνει μέχρι τώρα από ό,τι φαίνεται σε ορισμένες περιπτώσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο, όπως είπα, με έχει απασχολήσει πολύ. Το έχω συστήσει και με πολίτες στην Τσεχία. Απασχολεί πολύ τον κόσμο. Και άρα ερωτώ, εάν με αυτές τις μικρές μη κυβερνητικέ οργανώσεις έχετε την ευκαιρία καταρχάς να συνεργάζεστε, και ιδιαίτερα τι είδου δυνατότητε για εμβάθυνση αυτών των σχέσεων και τη συνεργασία βλέπετε. Ευχαριστώ κυρία Παρβάνοβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα ήθελα να σας συγχαρώ για τις, ε, καταρχάς για την ε, πρωτοβουλία, δεύτερον και για το μεγάλο θάρρος και την παρουσία που επιδεικνύεται προς, παρουσιάζοντας τα θέματα αυτά από κοινού. και τα αποτελέσματα της μελέτης που θα μας παρουσιάσετε. Υπάρχουν πολλές μελέτες από ό,τι φαίνεται, ανα, όχι μόνο την Ευρώπη αλλά και ανά ολόκληρο τον κόσμο, που μπορεί να μας δείξουν ε, σε, μεγάλο, σε μεγάλη έκταση την ενδοοικογενειακή βία και κυρίως τη μεγάλη διάχυσή της σε όλη την κοινωνία. Από αυτές τις μελέτες λοιπόν και από την χρήση τους για στόχους νομοπαραγωγικούς και κυρίως νομοπαραγωγική διαδικασία κυρίως σε θέματα πολύ ευαίσθητα όπως το ποινικό δίκαιο που μας απασχολούν στην Επιτροπή μας σε συνεργασία και με άλλους εισηγητές ε, στο νομοθετικό πακέτο για την προσοχή των θυμάτων την κυρία Χιμένα σαν προκειμένο βλέπουμε ότι οι θεσμοί σε όλα τα κράτη-μέλη, επίσημοι θεσμοί δείχνουν μια, ε, ε, κάποια επιφυλακτικότητα και δισταγμό απέναντί μας. Και πάνω απ' όλα γιατί αμφισβητείται η μεθοδολογία με βάση την οποία γίνεται η μέτρηση του, της έκτασης και του βαθμού της ενδοοικογενειακής βίας. Είναι αξιόπιστες οι δηλώσεις, οι καταγραφές, είναι ενδεχομένως συγκινησιακά φορτισμένες, υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία, πώς μπορούμε να κάνουμε δηλαδή μια ουσιαστική διάγνωση, διότι χωρίς αυτή δεν μπορούμε να έχουμε ούτε πρόληψη στοιχεία, ούτε και εντοπισμό των όποιων κενών στην ομοθεσία ε, θα έπρεπε να καλυφθούν ε, ώστε να προσφερθούν και οι πραγματικές, ε, πραγματικά απαραίτητες υπηρεσίες. Γι' αυτό λοιπόν και πιστεύω ότι είναι πολύ καλό εάν μια μελέτη όπως η δική σας μπορούσε να θεσμοθετηθεί και να αναγνωριστεί τυπικά από την Επιτροπή ώστε να αποτελέσει πηγή αναφοράς Επίσης και με τα εφιστάμενα δεδομένα, με τα στοιχεία που έχουμε στη θέση μας, είναι πολύ δύσκολο να διαπιστώσει κανείς γιατί και σε ποιες περιπτώσεις δεν καταγράφεται, δεν καταγγέλλεται η ενδοοικογενειακή βία ή ακόμα και αν καταγγελθεί γιατί οι γυναίκες παραμένουν θύματα, ε, στιγματίζονται δηλαδή ή έχουν τον κίνδυνο του ε, στίγματος, του θύματος ή γιατί δεν υπάρχει επαρκές σύστημα προστασίας όχι μόνο πρόληψης αλλά και προστασίας των θυμάτων της ενδοκιογενειακής βίας. Αυτά όλα τα στοιχεία λοιπόν θέλαμε να δούμε. Πώς οι υπηρεσίες χρειάζεται ενδεχομένω να προσαρμοστούν ώστε όχι μόνο να καταγράφουν κάθε στοιχείο σωστά, αλλά και να το καταγράφουν κατά τρόπο ουδέτερο, ώστε να μην ε, ε, εισάγονται διακρίσεις κριτική μεταχείριση. Ενδιαφέρον επίσης θα ήταν να γνωρίζουμε τι είδους κατάρτιση, εξειδίκευση ή με τι συστατικά εξειδίκευση θα πρέπει τα κράτη-μέλη να επιδιώξουν, να παρακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία. σε κάθε επίπεδο, μέχρι και το δικαστικό, αλλά και στη συνεργασία με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, διότι η πρόταση για εξειδίκευση, κατάρτιση εξειδικευμένη είναι πολύ διαδεδομένη, αλλά δεν αναφέρεται συγκεκριμένα ποιον θα πρέπει να στοχεύει, με τι περιεχόμενο, με τι αποτέλεσμα και σε τι ιδιαίτερα θα πρέπει να δοθεί ε, προσοχή. Όλα αυτά λοιπόν είναι πιστεύω στοιχεία που θα πρέπει που τον κόπο να διερευνήσουμε. Εν τέλει, Θα ήθελα συγκριτικά δεδομένα μεταξύ κρατών μελών. Και επίσης όταν μιλούμε για βία με βάση το φύλλο, ε, πολύ ενδιαφέρον είναι να δούμε και στοιχεία με βάση με μια ε, κατανομή αναεθνότητα ή ομάδα μειονοτική ή ιδιαίτερος ε, μετανάστες. Γιατί εκεί βλέπουμε, σε αυτές τις ομάδες κυρίως βλέπουμε, ότι συνεχίζονται αυτές οι πρακτικές και επίσης ε, εξακολουθούν να συγκαλύπτονται αυτές οι πρακτικές και να μην καταγγέλλονται. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παπαδοπούλου. Yes. Thank you very much. Actually, I... Σας ευχαριστώ. Και εγώ στην ίδια γραμμή με τη συνάδελφο θα θέλω να μιλήσω. Είναι πολλές, ε, πολλά τα χρόνια που συζητούμε για ουσιαστικές ε, και αξιόπιτες στατιστικές στο Συμβούλιο της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια ε, είχαν θεσπιστεί δείκτες 7 συνολικά με τη δυνατότητα για συγκρίσιμα στοιχεία μεταξύ κρατών μελών στο θέμα της βίας εις βάρος των γυναικών. Τώρα μας μιλάτε για 13 δείκτες και με... Ε, οφείλω να ομολογήσω ότι είμαι μπερδεμένη κάπως μου εξηγείτε παρακαλώ ποια είναι η διαφορά μεταξύ των 13 δικών σα και των 7 του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πρώτη ερώτηση. Και δεύτερον, για την Κύπρο. Είπατε ότι κατά τη διάρκεια της Προεδρίας θα έχετε συνεργασία για συλλογή στοιχείων που θα μπορούσε να αξιοποιήσει η Κυπριακή Προεδρία. Θα μπορούσατε να δώσετε πιο πολλά στοιχεία, παρακαλώ, για το θέμα αυτό. Καθώς είμαι Κυπρία, μπορώ να γνωρίζω ότι η κρατική μηχανή θέλει να έχει αξιόπιστες στατιστικές με πραγματικά γεγονότα, στηρισμένα σε πραγματικά γεγονότα. Είμαστε από τους πρώτους που είπαμε ότι εισάγουμε νομοθεσία από το Συμβούλιο της Ευρώπης, από τις πρώτες ε, χώρες, αλλά και από την, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, νομοθεσία που καταδικάζει την βία εις βάρος των γυναικών. Από την άλλη, δεν γίνεται λόγος επαρκής για την θέση του θύματος και το στεγματισμό του. Ε, και δεν έχουμε επαρκή στοιχεία. Γι' αυτό λοιπόν συμφωνώ με τη συνάδελφο ότι για να συλλεγούν αξιόπιστα στοιχεία θα πρέπει να βοηθήσουμε τις γυναίκες να ε, διαρρήξουν το κύκλο της σιωπή. Κάτι το οποίο δεν έχουμε επιτύχει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και έτσι Εάν ε, δεν μπορέσουμε να πείσουμε τη γυναίκα να φτάσει μέχρι την αστυνομία και να καταθέσει μήνυση κατά του θήτη, εάν δεν υπάρξει καταγγελία, πώς μπορούμε να έχουμε στοιχεία, πώς μπορούμε δηλαδή να ε, έχουμε και συλλογή στοιχείων και να πείσουμε το θύμα να μιλήσει. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είχε νομίζω επιτυχημένα ε, ευαισθητοποιήσει πριν από μερικά χρόνια σε μια εκστρατεία που είχε ξεκινήσει το κοινό. Αλλά δυστυχώ, δεν μπορέσαμε να επιτύχουμε αυτό, δηλαδή το να ε, καταγγέλουν οι γυναίκε θύματα τη ενδοοικογενειακή βία. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. σα δώσω και το λόγο για να απαντήσετε, έχω ακόμα δύο ερωτήσει. Κυρία Τόμσεν πρώτα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ για την πολύ καλή δουλειά που κάνετε. Είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον ότι η κατάσταση στα κράτη-μέλη εξελίσσεται. Θα ήθελα όμως ε, να γνωρίζω και αν τα διαφορετικά επίπεδα στατιστική στα κράτη-μέλη ή καταγγελίας στην αστυνομία της ενδοοικογενειακής βίας συνεχίζουν επίσης. Κάπου είχα διαβάσει ότι καταγγέλλονταν, ε, ότι θεωρούνταν μάλλον όσο πιο βίαιοι, οι πιο βίαιοι σύζυγοι οι Βρετανοί από την Ευρώπη των 15. Αλλά από την άλλη αυτό εξηγήθηκε και από το γεγονό ότι ήταν πιο πολλέ οι καταγγελίε ει βάρο των συζύγων από τι ε, συζύγου θύματα. Επομένω, πώ σταθμίζετε αυτά τα στοιχεία και πώ μπορείτε να έχετε επαρκή στοιχεία ώστε να ε, διαγνώσετε σωστά την εικόνα στα διάφορα κράτη-μέλη. Επίσης, Ποιε είναι οι δυσκολίε που θα αντιμετωπίσει μπροστά τη μια γυναίκα στον δρόμο προ το αστυνομικό τμήμα για την καταγγελία και ποια μπορεί να είναι η βέλτιστη πρακτική για τον περιορισμό τη βία. Η Ισπανία, παραδείγματι, η οποία έχει κάνει τις πιο πολλές προσπάθειες από όλες τις χώρες της Ευρώπης, διατηρεί ακόμη υψηλό τον αριθμό των θυμάτων των γυναικών, εκείνων που χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο λόγω της ενδοικογενειακής βίας. Τα δε άσυλα ή χώροι υποδοχής για γυναίκες και παιδιά θα ήθελα να γνωρίζω ακριβώς τι στοιχεία έχετε, γιατί βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά. Και μην ξεχνάμε ότι καλό θα είναι να δίνετε βέβαια και η σχετική θεραπεία στους άντρες, αλλά μην ξεχνάμε και τις γυναίκες. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τελευταία ερώτηση, η κυρία Χιμένες. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να χάσουμε την ευκαιρία του να συγχαρούμε για το έργο που επετέλεσε και για την εισήγησή της την προσκεκλημένη μας. Εγώ από την εμπειρία μου ως εισηγήτρια, ως εισηγήτρια, ως κοιόδης εισηγήτρια στην έκθεση κυρία Βένσον για την βία μεταξύ των δύο φίλων ε, και πρέπει να σας πω ότι ήταν ε, έκθεση που συν... τη Γενική Συνένεση και έχουμε επίσης τώρα το θέμα της προστασίας των θυμάτων, τον έχουμε και κάποιον φορέα, έχουμε την έκθεση Παρβάνοβα, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσουμε την υποστήριξη όλων των θυμάτων. Των θυμάτων της βίας και οπότε αυτό το οποίο ό,τι ότι έχει σχέση με στατιστικές από ό,τι φαίνεται χαρακτηρίζεται από κάποια παθητική αμυντική πολιτική και ότι τα κράτη-μέλη έχουν πρόβλημα όσον αφορά το να κοινοποιήσουν τα δεδομένα που στη διάθεσή τους. Επίσης, άλλο πρόβλημα είναι ότι από φόβο ή από το ότι θα τις κατηγορήσουν οι γυναίκες δεν καταγγέλουν τα φαινόμενα της βίας. Και συγκεκριμένα στην Ισπανία ουσιαστικά έχουμε ένα 20% των καταγγελιών που έρχονται από την ε, αστυνομία και όχι από το ίδιο το θύμα. Και εμείς με το ρόλο που έχουμε ως νομοθέτες προσπαθούμε επί τη βάση των σημαντικών αυτοσταστικών να νομοθετήσουμε. Επομένως χρειαζόμαστε την βοήθειά σας, την αρρωγή σας και φυσικά και μας ε, περιμένουν πώς και πώς να ακούσουμε τη γνώμη σας, πώς μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε τώρα, από, από πλευρά κάποιου συμπεράσματο και δευτερολογία, να δώσουμε τον λόγο στι δύο συγκήτρες με όποια σειρά θέλουμε να λάβουν τον λόγο. Να μιλήσουν. Εσύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω ό,τι μπορώ, ούτω ώστε να καλύψω όσα έχουν ερωτηθεί. Πρώτη ερώτηση. Ο Οργανισμός Τελευταίων Δικαιωμάτων έχει μια πλατφόρμα δικαιωμάτων και εκεί έχουμε 350 φορείς αλλά και για την έρευνα αυτή συνεργαστήκαμε πάρα πολύ στενά με την Wave οι οποίοι επίσης μας έδωσαν πληροφορίες για αυτό τα άσυλα καταφύγια γυναικών στα κράτη-μέλη και εμεί προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε το ότι κατά αυτή την διαρκή του επινέρου των 40.000 γυναικών να αναζητούσαν ε, να δούμε αν είχε αναζητηθεί εκεί η βοήθεια. Ήταν κομμάτι αυτό της έρευνας η συνεργασία με τις μη κυβερνικές οργανώσεις και να δούμε Εάν μπορούν τα αποτελέσματα να φτάσουν εκεί που τα χρειάζονται περισσότερο τώρα. Επίση τα αποτελέσματα δείχνουν το αν ξέρουν για την υπαρξή των οργανώσεων οι γυναίκε. Του δείξαμε ένα κατάλογο και ρωτήσαμε αν έχουν ακούσει. Βέβαια, από όλη χρηματοδότηση πολλέ φορέ δεν είναι γνωστή η ύπαρξη αυτών των οργανώσεων. Οπότε έτσι χαρτογραφούμε το τοπίο με κάθε τέτοια έρευνα Ξεκινώ όμως με κάποιο τυχαίο δείγμα για το τι ξέρουν αυτές οι γυναίκες και για το εάν αναφέρουν σχετικά στην αστυνομία, σε για οργανώσει, στην οικογένεια, στους φίλους τους. Επομένω, αυτή είναι η απάντηση ότι ναι, συνεργαζόμαστε με συγκεκριμένες οργανώσει και επομένω είναι χαρά μας το να είναι χρήσιμο το πλούσμα της έρευνα στι στις μη κυβερνικές οργανώσεις. Και αυτό αφορά όλους τους εμπλεκομένους, όλου όσου ασχολούνται με το φαινόμενο αυτό τη βία. Επίση, έχουμε και άλλε έρευνε στο Νέο Βασίλειο και αλλού. η κυρία Παρβάνοβα το ανέφερε και χρησιμοποιούν τι έρευνε για την νομοθεσία και δια... τυπώνται πάντω κάποιε επικρίσει. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ των στατιστικών τη διοίκηση, τη ποινική δικαιοσύνη, την άλλη μεριά, γιατί πάντα υπάρχει διαφορά γιατί διαφέρει το ποινικό δίκαιο τι και πώς το τα σε κάθε μέλος. Όταν έχω μια έρευνα για τα θύματα βίας, όπως τα δικά μας, τότε προκύπτει συγκρισιμότητα. Χρησιμοποιείται ακριβώς η ίδια δειγματοληψία, ακριβώς το ίδιο ερωτηματολόγιο, μεταφρασμένε διαφορετικές γλώσσες και άρα είμαστε όσο γίνεται πιο συγκρίσιμοι όσο πιο κοντά γίνεται με τις στατιστικές της επίσημης της ποινικής δικαιοσύνης. Νομίζω η κυρία Τόμσον είπε για το νούμερο Βασίλειο. Και εκεί προκύπτουν πάρα πολλές τέτοιε περιπτώσεις και εκεί ενθαρρύνεται, υπάρχει δυνατότητα της καταγγελίας. Αν όμω βάλουμε και συγκρίνουμε δίπλα τα στοιχεία ε, του Οργανισμού Θεμελιών Δικαιωμάτων. Θα δούμε μόνο ποια είναι τα επισημαστικά και τι μας λένε στην έρευνα. Θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει το εξή. Η Άγκη ασχολείται με αυτά τα στοιχεία και επισημαίνει ποια είναι τα προβλήματα της συγκρισιμότητας. Εμείς συνεργαζόμαστε με την Eurostat. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι ξέρουν για την μελέτη την έρευνα και έτσι τον προλέρουμε το έδαφος για την επόμενη έρευνα. Γιατί υπάρχουν κάποια στοιχεία που έχουν, αλλά δεν είναι αρκετά. Οπότε, τα δικά μας δεδομένα βασίζονται σε κάποια κλασική, σε κάποια αποδεκτή από τους μεθοδολογία και έχουμε πολλούς συμπεριγνώμες που το εξασφαλίζουν. και κάτι άλλο τρόπο αναφέρθηκε όσον αφορά την κατάρτιση, εκπαίδευση. Αυτό το οποίο εμείς θέλουμε να βγει από το αποτελέσμα τη έρευνα είναι να χρησιμοποιηθεί από πολλούς σημαντικούς παράγοντες ε, για την ε, κατάρτιση, εκπαίδευση, στην χώρα τη απασχόληση της αστυνομία και έχουμε δημοσιεύσει διάφορες μελέτες. Μία άλλη που έλεγε όταν Ευρωπαϊκή Ένωση Μίδας Εκεί είχαμε 23.000 περίπου ε, μετανάστες εθνοτικών ομάδων και αυτό χρησιμοποιήθηκε σε ένα εγχειρίδιο για την αστυνομία, από την αστυνομία επίσης. Άρα να, αν καταλήξει κάποιο εγχειρίδιο όλο μας το έργο, αυτό θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Όμως θέλουμε οι εμπλεκόμενοι να μας βοηθήσουν και έτσι να φροντίσουμε εμείς για την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων. Τώρα, όσον αφορά για κάποια για τους ε, μετανάστες που δεν έχουν καταγραφεί και για κάποια εθνοτικά ευαίσθητα στοιχεία. Η έρευνα αυτών, επειδή πολλές φορές είναι παράνομη ή μη καταγεγραμμένη, το ε, παρουσιάζει προβλήματα στην ε, δειγματοληψία. Κρύβονται, φοβούνται, φοβούνται με τους, με τους διώξαν τη χώρα. Όμως πέρσι δημοσιεύσαμε τρεις τέτοιες εκθέσεις για για αυτούς τους λάθρομετανάστες, τους πάνω μετανάστες ε, και τις γυναίκες που δουλεύουν ε, και βοηθάνε στα νοικοκυριά, στα σπίτια και ε, για τη βία κατά αυτών. Αλλά όπως προείπαμε, μια έρευνα τέτοια μετακαλύψει τα καλύψει όλα. Τώρα αφορά τα κριτήρια δείκτες, έχουν πολλούς διαφορετικούς δείκτες. Όμως δεν χρησιμοποιούνται τα κριτήρια του ΟΗΕ. Αυτή τη διαδικασία διάρθρωση όπως ονομάζεται και άλλωστε αυτοί οι δείκτες χρησιμοποιούν και για, χρησιμεύουν για άλλες έρευνες όπως ασία δεδομένων κλπ. Θα προσπαθήσω κι εγώ να να απαντήσω. Καταρχήν, ε, ναι, και πολύ σχεδόν το Ινστιτούτο συνεργάζεται με τις ΜΚΟ και τους διάφορους stakeholders, με τα διάφορα διαφορεμένα μέρη, με πολλαπλούς τρόπους. Καταρχήν, στη μελέτη για την υποστήριξη των θυμάτων θα συμμετέχουν και ΜΚΟ στη συλλογή των δεδομένων και θα πω δύο λόγια παραπάνω για το πώς, γιατί δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσω για τη μεθοδολογία της μελέτης. Ε, οι ΜΚΟ θα παρέχουν τα δεδομένα Δεύτερον, να συμμετέχουν γιατί μας παρέχουν εμπειρογνωμοσύνη. Το αναφέρατε ήδη τα δίκτυα κατά των ε, γυναικών και το European Women Lobby είναι οργανώσεις ε, και έχουμε και οργανώσεις ε, σε επίπεδο κράτους μέλους που συμμετέχουν στο δικό μας έργο. Το τρίτο είναι ότι το Ινστιτούτο πρόσφατα ολοκλήρωσε ένα πολύ μεγάλο έργο χαρτογράφηση των ενδιαφερομένων μερών έχουμε 50.000 καταχωρήσεις εκεί, διάφορες οργανώσεις που εργάζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών και αυτή η βάση δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας για την ανταλλαγή πληροφοριών, για την αλληλοενδυνάμωση, αν ζητούν εταίρους για ε, τα project τους ε, και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν αυτές οι διαφορετικές βάσεις δεδομένων και πλατφόρμα θα εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς γιατί μία από τις εντολές του Ινστιτούτου είναι να αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο για την ισότητα των δύο φύλων. Γι' αυτό έχουμε κάνει αυτή τη χαρτογράφηση και έχουμε ε, αυτή την βάση δεδομένων για τα ενδιαφερόμενα μέρη από τις διάφορες χώρες και φυσικό οι NGO πολυπλασιάζουν, οι μη κυβερνητικές οργανώσει πολυπλασιάζουν τα δεδομένα γιατί μα βοηθούν να διαδώσουμε τα αποτελεσματά μας στους τελικούς χρήστες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συγκρισιμότητα των δεδομένων, και εδώ ίσως θα πω δύο λόγια για τη μεθοδολογία σε ό,τι αφορά τη μελέτη υποστήριξη των θυμάτων που θελοποιήσουμε σε κάθε χώρα. Θα έχουμε τρει παροχού δεδομένων, εκπρόσωποι της κυβέρνηση, των ΜΚΟ και από το ακαδημαϊκό κύκλο, που θα μα δώσουν δεδομένα για τι διαθέσιμε υπηρεσίε σε κάθε χώρα έχουμε 13 υποδείκτες, δηλαδή 13 είδη υπηρεσιών που θα μας βοηθήσουν να χαρτογραφήσουμε. Και εντός αυτού θα επικεντρωθούμε σε γενικές υπηρεσίες και σε ειδικέ υπηρεσίες. Με τις ειδικέ υπηρεσίες εννοούμε αυτές που πραγματικά ε, συγκεντρώνουν εμπειρογνωμοσύνη και ειδική γνώση το πώς θα εργαστούμε με τις γυναίκες ε, και εφαρμόζουν την προσέγγιση του φύλου ε, στην εργασία αυτή. Και τι το κάνουμε αυτό, το κάνουμε για να δούμε εάν είναι σκόπιμο ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών. Και ένα από τα σημεία εστίαση ε, δεν θα είναι μόνο τα αριθμητικά στοιχεία, δηλαδή να δούμε πόσε υπηρεσίε έχουμε, αλλά να αξιολογήσουμε και την ποιότητα των υπηρεσιών. Και εντό αυτού θα θέλαμε να δούμε ποια είναι τα εμπόδια που εμποδίζουν, ποια είναι τα εμποδία, γιατί οι γυναίκε δεν επιλέγουν κάποιε υπηρεσίε, γιατί δεν πηγαίνουν στην αστυνομία να καταγγείλουν, ε, ποια είναι τα προβλήματα ε, με ε, Οργανισμού οργανισμούς περίθαλψη περίθαλψης ε, και να σα πω, έχουμε στοχεύουμε πάρα πολύ στο πώς θα συλλέξουμε τις βελτικές πρακτικές και πώς το εσωτερικό των οργανισμών θα αντιμετωπίσουμε τα θύματα προκειμένου να καταστούν ε, ορατές ε, αυτές οι πρακτικές και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις γυναίκες θύματα. Όμως τα πρωτογενή δεδομένα θα είναι συγκρίσιμα. Θα είμαστε σε θέση να τα συγκρίνουμε αυτά τα δεδομένα γιατί για τις εκθέσεις των προεδριών υιοθετούμε εφαρμόζουμε την ίδια μεθοδολογία σε όλες τις χώρες και σκοπεύουμε στο να έχουμε συγκρίσιμα δεδομένα. Ε, βέβαια υπάρχουν και κάποιες επιφυλάξεις και θα τις ε, Τώρα, ρωτήσατε για τους 7 και τους 13 δείκτες. Έχουμε 7 δείκτες που έχουν εγκριθεί, ένας από αυτούς είναι η υποστήριξη των δημάτων. Και για την υποστήριξη των δημάτων έχουμε 13 υποδείκτες. Και τώρα θα ήθελα να πω και λίγα λόγια για τις εθνοτικές μειονότητες ε, ε, ένας από τους υποδείκτες ε, είναι οι υπηρεσίες που παρέχονται σε ευάλωτες ομάδες γυναικών. Όταν λέμε ευάλωτες ομάδες εννοούμε εθνοτικές μειονότητες ή πολιτιστικές μειονότητες. Η Ρωμά, παραδείγματο χάρη, οι γυναίκες Ρωμά είναι, δεν είναι εθνοτική μειονότητα ή οι γυναίκες LGBT, οι ομοφιλόφιλες, οι ε, γυναίκες. Θα δούμε δηλαδή πώς μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσία σε αυτές τις ευάλωτες ομάδες γυναικών. Και τώρα η εστίαση στους δράστες και στα άσυλα. Σε όλο και περισσότερες χώρες ε, βλέπουμε να γίνεται μεγαλύτερη συζήτηση για τις εντολές προστοσίας, δηλαδή πώς θα απομακρυνθεί ο φίτης ε, από το σπίτι θέλουμε να καταστήσουμε να προβάλλουμε αυτό το θέμα, να το καταστήσουμε ορατό. Τα άσυλα είναι σημαντικά, αλλά δεν αποτελούν τη λύση στο πρόβλημα. Και πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι με τους δράστες και το πρόγραμμα απομάκρυνσης των δραστών επίσης θα πρέπει να λειτουργεί. Γιατί όταν οι γυναίκες πρέπει να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, ε, υφίστανται δευτερογενή θυματοποίηση θυματοποιούνται για δεύτερη φορά. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταστήσουμε αυτό ορατό. Σας ευχαριστώ. Uh, I'm not speak Swedish. Θα μιλήσω πάλι σουηδικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τις δύο ομιλήτριες που ήρθαν εδώ να μας ενημερώσουν για τη δουλειά τους. Μπορεί καμιά φορά να δίνεται η εντύπωση ότι στα στατιστικά και τα δεδομένα είναι μια δουλειά στεγνή, αλλά όχι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα, κυρίως αν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετική αξιολόγηση, στάθμιση των δεδομένων αυτών και πάνω απ' όλα εάν παρουσιάζονται, όπως έγινε εδώ, τα στοιχεία με την κωδικοποίησή τους και ε, βεβαίως με την ε, ενημέρωση για το πώς θα μπορούσαμε εμείς να αξιοποιήσουμε τα στοιχεία αυτά πιο πρακτικά στη δουλειά μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν θερμά. Τώρα. προχωρήσουμε τώρα στο πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και την ε, καινοτομία. Παρακαλώ. Ανάλυσα την πρόταση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για τη δημιουργία ενός προγράμματος ε, για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία και πρόσεξα ότι σε αυτό το σχέδιο κειμένου λείπει η πτυχή του φύλου και δεν αναφέρεται ποτέ το θέμα των ίσων ευκαιριών το πρόγραμμα θα πρέπει να ακολουθήσει έναν από τους κύριους στόχους που είναι η ενίσχυση της παρουσίας της απασχόλησης των γυναικών στην αγορά εργασίας και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των γυναικών για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε το πώς θα συμφιλιώσουν την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή. Παρουσίασα λοιπόν 15 τροπολογίες σε αυτή την πρόταση κανονισμού το πρόγραμμα θέλει να συνεισφέρει ε, στην, ε, υλοποίηση της στρατηγικής του 2020 ε, υλοποιώντας και σημαντικούς στόχους για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ αυτών η πρόθεση ενός υψηλού επίπεδου πασχόλησης η εγγύηση μιας κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, επαρκούς κοινωνικής προστασίας, βελτίωση των εργασιακών συνθήκων και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της ανέχειας. Πρόκειται για στόχους ε, στους οποίους πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από την πολιτική που ασχολείται με την ισότητα των φύλων και θα ήθελα λοιπόν να αναλύσω κάποιες από αυτές τις τροπολογίες που παρουσίασα και κατόπιν να βελτιώσω αυτή τη γνωμοδότηση και με τη συνεισφορά των συναδέλφων. Τροπολογία 1 εδώ δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην πρόθεση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των γυναικών, δεδομένου ότι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο μία στι δέκα γυναίκες είναι επιχειρηματίας. Ενώ ε, για τους άνδρες ισχύει ένα στους τέσσερις. Έτσι λοιπόν... Ε, πρέπει να ευνοήσουμε την πρόσβαση των γυναικών στην μικροπίστωση. Τροπολογία υπεριθμών 5. Εδώ δίνουμε έμφαση στη δημιουργία θέσεων απασχόληση που να δίνουν τη δυνατότητα στους εργαζομένου να πετύχουν υγιή ισορροπία μεταξύ επαγγελματική και ιδιωτική ζωή. και για τη χρηματοδότηση των μελλοντικών ε, έργων μέσω αυτού του προγραμμάτος, μέσω της τροπολογία 8, έχω ζητήσει μία προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη το φύλλο πάντοτε, ε, για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις κατά των γυναικών ε, στο χώρο της εργασίας. Κατόπιν ε, επικεντρώνομαι στο άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού αυτού στις άμεσες δράσεις για την προώθηση της κοινωνικότητας των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, όπως πολλάκις υπόθηκε, δίνουμε μεγάλη σημασία στο να ευνοήσουμε τη θέση της γυναίκας στον χώρο της εργασίας για να μπορέσουμε να βγούμε και από τη σημερινή οικονομική κρίση που πλήττει πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση. Είμαι λοιπόν πεπισμένη για το στρατηγικό ρόλο που μπορεί να έχει η γυναίκα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο τροποποίησα την τροπολογία 10 ε, βάζοντας και τον ε, ειδικό κατάλογο εργαζομένων όπως ε, παραδείγματο χάρη έχουμε τις γυναίκες και τους άνδρες που εργαζόνται σε μερική απασχόληση και έχουν αναλάβει να φροντίζουν κάποιον άρρωστο ή άλλες ομάδες εργαζομένων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα της συμπληρωματικότητας ε, του προγράμματος αυτό με άλλες δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω την τροπολογία 11 για το άρθρο 8 παράγραφος 1 για την ισότητα των φύλων μεταξύ των ε, διάφορων τομέων δράσης της Επαγγελματικής Ένωσης, ε, εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, υγεία, έρευνα και καινοτομία. Για ε, μια ακόμη φορά λοιπόν ε, έλειπε η, η πτυχή του φίλου στο πρόγραμμα αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα τις διετής εκθέσεις παρακολούθησης, ε, που η Κομισιόν διαβιβάζει στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Η τροπολογία 12, όπως είναι απαραίτητο, αναφέρει ότι στις εκθέσεις αυτές πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ακόμη περισσότερο οι αρχές της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών για τι ενσωμάτωση τη διάσταση του φύλου σε ό,τι αφορά κυρίως το θέμα της μη εισαγωγή διακρίσεων. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση, ωστόσο δεν ε, μπορέσα λοιπόν ε, να έχω ιδιαίτερα μακροσκελείς τροπολογίες. Έπρεπε να σεβαστώ τους κανόνες ε, για να μπορέσω να συντάξω τη γνωμοδότηση αυτή. Όμως οι συνάδελφοι σίγουρα θα μπορούν να μου δώσουν χρήσιμες πληροφορίες, είμαι σίγουρη θα μου πούν ε, πού μπορεί να βελτιωθεί αυτό το σημαντικό σχέδιο κανονισμού, γιατί μιλάμε για ένα μελλοντικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορώ να πω ότι στο σημερινό πλαίσιο γίνεται τόσος λόγος για την κοινοτομία και την αλλαγή. Έτσι λοιπόν πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτή τη γνωμοδότηση. Πραγματικά πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Eh, ευχαριστώ. Και τώρα... επιτρέψτε μου να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, κυρία Ζήμπα. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή. Εμείς θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι αυτό το πρόγραμμα είναι πολύ σημαντικό ιδίως ε, λόγω της συγκυρίας ε, στην οποία βρισκόμαστε, ως συνέπεια της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, οι γυναίκες πλήττονται ακόμη περισσότερο ε, στον τομέα της απασχόλησης, πολύ περισσότερο από τους άνδρες και ιδίως μέσω της μείωσης των μισθών τους μέσω της επισφαλούς απασχόλησης. Ξέρουμε ότι οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο από αυτή την επιτυχή, από αυτό το φαινόμενο και επίσης και από την ανεργία. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτό το πρόγραμμα μπορεί να έχει ένα, θεμελιώδες, ε, ένα θεμελιώδη ρόλο ε, και αναφέρομαι στο θέμα της μικροχρηματοδότησης και εμείς ε, ως σύγκριτες της πρότασης αυτής στην Επιτροπή προτείνουμε ο φορέας της μικροπίστωσης να αυξηθεί δηλαδή μικροπιστήση να αυξηθεί σε σχέση με τις άλλες δύο συνιστώσεις ε, και θεωρούμε ότι και οι άλλες δύο συνιστώσεις ε, είναι σημαντικές, αλλά εμείς θεωρούμε ότι η μικροχρηματοδότηση είναι η συνιστώσα η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο πρακτικά αποτελέσματα ως προς την δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν Συμφωνώ όμως ε, λέγονται και θέλουμε να πούμε ότι θα παρουσιάσουμε προτάσεις προκειμένου το θέμα της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων να λαμβάνεται παρκώς υπόψη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στο στριτογενή τομέα και στη λεγόμενη κοινωνική οικονομία όπου έχουμε τομείς όπως ε, ε, οι κοπερατίβες, ε, οι οργανισμοί αλληλοβοήθειας και εμείς ε, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικοί αυτοί οι οργανισμοί γιατί υπάρχει αναδιανομή των ε, κερδών στους ε, εταίρους που συμμετέχουν σε αυτές τις επαγγελματικές ενώσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπιλμπάου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την κυρία Ματέρα για τις εξηγήσεις που μας έδωσε. Καταρχήν, να πω ότι η πρόταση κανονισμού που παρουσιάστηκε από την ε, Επιτροπή ε, έχει να κάνει με την ε, εκτέλεση των στόχων του προγράμματος του 2020. Αναφέρεται στο πρόγκριστο, στο Γιούρες, στην μικροπίστωση, στη μικροχρηματοδότηση και λέγεται ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη δύο πράγματα για την επιτεύξη των στόχων. Καταρχήν, την πρόθεση της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων, αλλά ε, παρόλα αυτά μόνο σε αυτή την παράγραφο αναφέρεται η ισότητα των δύο φύλων ε, και σε κανένα άρθρο δεν αναφέρεται πώς θα υλοποιηθεί αυτή η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά πρέπει να εκτελεστούν τα προγράμματα αυτά. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι έχουμε ε, έλλειψη ενός από τους στόχους που θέτει η ίδια η Κομισιόν. Προκειμένου να καθορίσουμε τη δική μας θέση, να πω ότι συμφωνούμε με τις τροπολογίες, αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάμε παραπέρα, γιατί ο τίτλος αυτής της πρωτοβουλίας είναι «Κοινωνική αλλαγή και καινοτομία» και νομίζω ότι μπορούμε να εισαγαγούμε τουλάχιστον νομίζω από τη δική μας ομάδα, αυτό θα κάνουμε, θα καταθέσουμε τροπολογίες προκειμένου ε, η συμμετοχή των γυναικών ε, στον ε, στο χώρο της εργασίας και η οικοδόμηση της ισότητας ισούται με την κοινωνική αλλαγή και αυτό μπορεί να μας επιτρέψει να έχουμε έναν ακόμη παράγοντα για να βγούμε από την οικονομική κρίση. Ακριβώς βάσει και των στοιχείων που έχουμε από όλες τις έρευνες, οι Ευρωπαίες έχουν καλύτερη μόρφωση και κατάρτιση. Οι γυναίκες στην Ευρώπη παράγουν καλύτερα αποτελέσματα ε, στον τομέα της οργάνωσης, ε, είτε στις επιχειρήσεις, ε, είτε σε άλλες οργανώσεις, σε άλλους οργανισμούς. Έτσι λοιπόν θα παρουσιάσουμε τροπολογίες προκειμένου να ενισχύσουμε ε, τη συνεκτικότητα του τίτλου σε κάθε μία από τις πτυχές και τα προγράμματα και επειδή πιστεύουμε ότι η κοινωνική κοινοτομία πρέπει να πάει παραπέρα, πέρα από την επίτευξη της ισορροπίας ε, ε, μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δεν θέλουμε μόνο αυτό, αλλά μέσω τη ισότητας θέλουμε να έχουμε και κοινωνική καινοτομία και μέσω τη κοινωνική νομοθεσία να επέλθουν και μέτρα για, την, για το ξεπέρασμα τη κρίση. Και πιστεύουμε ότι η συμπερίληψη των γυναικών είναι ένας παράγοντα κλειδί για τη συγκυρία αυτή. Σα ευχαριστώ. Eh, Δεν βλέπω να ζητεί κανεί άλλο το λόγο. Ε, στρέφουμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλετε να λάβετε το λόγο. Υπάρχει πρόσωπος επιτροπής εδώ. Μάλιστα, καλώς. Τότε παρακαλώ την κυρία Ματία να λάβει το λόγο και πάλι για να κλείσουμε. Ευχαριστώ. Δεν έχω πολλά να προσθέσω στην παρουσίαση που έκανα προ λίγων λεπτών. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σημειώνω τα σχόλια των συναδέλφων γιατί και εμένα με εξέπληξε ότι ο τίτλος ε, δεν συνάδει με το κείμενο. Ε, όπως ε, είπε και η συνάδελφος η κυρία Μπιλμπάου, έτσι λοιπόν πρέπει να εργαστούμε στο να υπάρχει πραγματική ισότητα. Και περιμένω τις τροπολογίες και από τους συναδέλφους που δεν είναι παρούσες, γιατί είμαι σίγουρη ότι το θέμα αυτό είναι στρατηγική σημασία σε αυτή τη στιγμή, αλλά φυσικά και για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποτελέσει ε, μια σημαντική συνιστόσα. Eh, då vill jag bara annonsera att eh, det sista Καλώς, ευχαριστώ. Το μόνο που έχω να πω πλέον είναι ότι έχουμε για τι τροπολογίε ω προθεσμία της 2 Μαΐου, 5 το απόγευμα. Στι 13 του Μαΐου θα γίνει η ψηφοφορία στην Επιτροπή μα, 30 διορθώνουμε. Και στι 31 30-31 Μαΐου στην Επιτροπή Ψηφοφορία και Ολομέλεια τον Ιούλιο. Και έτσι ολοκληρώνεται το θέμα αυτό τη σημερινή διάταξη. Και τώρα πάμε στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατάληξη του κανονισμού υπαριθμών 1081-2006. Εδώ είχε προβλεφθεί ο κύριος Σιμάνσκι, ο συντάκτης, αλλά ε, κολλείεται σήμερα. Και έτσι παρακαλώ τον κύριο Βορζοβουζίτη να λάβει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είπατε πολύ σωστά. Είναι απόρρο, ο κύριο Σιμάνσκι, ζητεί συγγνώμη. Έχει ένα οικογενειακό λόγο σοβαρό που δεν μπορεί να έρθει, Ζητή συγγνώμη σας λοιπόν. Και με παρακαλεί να παρουσιάσω εγώ πολύ σύντομα την γνωμοδότησή του για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η τροποποίηση του κανονισμού είναι σημαντική. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία και στο ρόλο τη αρμόδια πολιτική, αλλά και στη λειτουργία του Ταμείου στι χώρε Ανατολική Ευρώπη, από την εποχή που ε, με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει σημαντικά περιορίσει τα προβλήματα και τις δυσκολίες σε κοινωνικό επίπεδο. Δηλαδή αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό κεφάλαιο για τις ε, χώρες, της περιοχές αυτές. Ε, βοηθά στην αντιμετώπιση τη κοινωνική κατάρτιση, ε, του κοινωνικού αποκλεισμού, ενίσχυση τη κατάρτιση και το καθεξής. Στο πλαίσιο λοιπόν τη πρόθεση κοινωνική ένταξη και τη καταπολέμηση τη φτώχεια, πρέπει να σημειωθεί ότι φυσικά πολύ να χορηγηθεί η στήριξη στι γυναίκε που βρίσκονται σε, μεγαλύτερη, σε δύσκολη επαγγελματική κατάσταση, δεδομένου ότι αυτέ διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο τη φτώχεια, καθώ και να στηριχθούν οι μονογονικέ οικογένειε και ιδιαίτερα οι μόνε μητέρε, με σκοπό να διευκολυνθεί ο συνδυασμό τη επαγγελματική και τη οικογενειακή ζωή. επίση, ευελιξία, ζητά ελαστικότερε διατάξει του κανονισμού που επιτρέπουν στα δεδομένα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν τα συγκεκριμένα δικά του κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα. Αυτό αφορά μεταξύ άλλων και του στοχευόμενου δικαιούχου του Ταμείου και το αίτημα ο κανονισμό να μην καθορίζει κάποιου περιορισμού. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Κυρία Χιμένας, παρακαλώ. Εκπροσωπώ την κυρία Σαμπρόσκα που απουσιάζει. Γιατί είχε μια ερώτηση. Ευχαριστεί λοιπόν τον κύριο Σιμάντση για τις προτάσεις του που ιδιαίτερα στοχεύουν τις πιο ευάλωτες ομάδες, γυναίκες δηλαδή, μονογονικές οικογένειες και το που κινδυνεύουν από τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ε, ιδιαίτερα λοιπόν αυτό έχει να κάνει και με τις ευθυγραμμίστικες και στις μακροχρόνιες θέσεις της ε, Επιτροπής μας αλλά και του ΕΛΚΑ. Ιδιαίτερα ο κίνδυνος του, της και του κοινωνικού αποκλεισμού πρέπει να αντιμετωπιστεί και ιδιαίτερα θα ήθελα να πω ότι συμμερίζομαι με τις ε, θέσεις του κυρίου Σιμάνσκι ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη, τα επιμέρου κρατη κράτη-μέλη να προσδιορίσουν τα, ποια είναι τα, ε, ποιες είναι οι περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες, γιατί δεν ισχύουν τα ίδια μέτρα και σταθμά παντού και ιδιαίτερα σε σχέση με τα παλαιότερα ή τα πιο πρόσφατα κράτη-μέλη. Έτσι θα μπορεί να καταστεί πιο αποτελεσματικό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Επίση, χαίρομαι που ο κύριο και σημαίνει ότι στην ποιότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών θα πρέπει να αναγνωρίζεται η διαφορά μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού βίου. Βλέπουμε ότι η οικογενειακή ζωή, τα παιδιά μπορεί να μετατραπούν σε παράγοντα Διάκριση ει βάρο όποιου τα φροντίζει για την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε πάνω απ' όλα λοιπόν. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Χάνιμπολ. Πρόεδρε ευχαριστώ. Θέλω να προσθέσω τα εξή. Κάποια στιγμή, σε λίγη ώρα, θα συζητήσουμε για τον προπολογισμό, οπότε θα πρέπει να το δούμε και αυτό το θέμα πώς πάει ως προς τον προπολογισμό και να μην ξεχνούμε τα θέματα αρμοδιότητά μα και το ότι δεν σταματάει ο αγώνα μα κατά τη διάκριση ει βάρο των γυναικών σε κάθε επίπεδο. Φυσικά και συμφωνώ με όλα όσα ε, ακούστηκαν σε σχέση με, με, με τη φτώχεια κλπ. Γιατί είναι αλήθεια ότι οι γυναίκε ε, υποφέρουν δυσανάλογα από την φτώχεια. Άρα θα πρέπει να συνεχιστεί χωρί σταματημό ο αγώνα. Συμφωνώ με όλα αυτά και επίσης θα πρέπει, όπως προελέχθη, να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε προσβασιμότητα και σε κάποια άλλα προγράμματα, τα οποία δεν τα συζητάμε εμεί εδώ, αλλά αλλά εν έχουν σχέση με τη δουλειά μας. Αποτελούν πηγές ενδιαφέροντος όπως το κοινωνικό ταμείο, οπότε Νομίζω ότι είναι αξιόλογη αυτή η έκθεση, είναι αξιόλογα στοιχεία. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Δεν ξέρω, δεν το λόγο ο συνάδελφος που προηγουμένως. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. νομίζω ότι έτσι φαίνεται πόσο σημαντικά θεωρούμε και θεωρείται όλα αυτά. Επίσης, επειδή είμαι και μέρος των προπολογισμών, σας επιβεβαιώνω ότι έχουμε πάρα πολλούς πόρους οι οποίοι προέρχονται από το Γενικό Ταμείο και φυσικά η Πολωνία έχει ωφεληθεί. Όλα όσα είπατε, πρόκειται να τα διαβάζω στον κύριο Σιμάνσκι και είμαι σίγουρος ότι θα ευχαριστεί πάρα πολύ με όλα αυτά που ακούστηκαν. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Τη Δευτέρα Μαΐου στις 5 το απόγευμα λίγη προθεσμία για υποβολή τροπολογιών. 30 Μαΐου θα ψηφίσουμε και επιστροφή Επιστροπή στι στις 10 Ιουνίου. Επομένως, τώρα προχωρούμε στο σημείο παριθμών 8 της διατάξεως. Γιατί το 7 θα το συζητήσουμε την Τρίτη. Άρα να βάλετε σε αυτό το σημείο. Πρόκειται τώρα για ανταλλαγή απόψεων του κ. Τζοβάνι, δηλαδή ασυγητή των προπολισμών του 2013. Όμως ο κύριος Λαδία δεν ήρθε ακόμη. Άρα να δώσουμε λόγο στην κυρία Χανίμπολ για να κάνει τη σχετική εισήγηση. Και θα πάρετε σκητάλη όταν έρθει ο κύριος Λαδία. Κυρία Χάνιμπολ. Ναι, φτάσαμε κάπως νωρίς σε αυτό το σημείο δυστυχώς, αλλά θα κάνω και εγώ ό,τι μπορώ. Και ίσως να μου ξαναδώσετε το λόγο αφού ακούσω τι έχει να μας πει ο κύριος Λαβία, γιατί έχει σημασία το θα πει. Το βασικό θέμα και η δυσκολία του προπολογισμό, κάτι περισσότερο από ό,τι άλλη χρονιά είναι ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την κρίση παντού, σε όλα τα κατημέρια. Λιτότητα παντού, περικοπές και όλες τις συνεπιές τους. Κανένας, κανένας δεν τη γλιτώνει. Άρα προφανώ θα πρέπει να θεωρηθεί από αυτή την οπτική γωνία. Θεωρείται ότι θα πρέπει ο προηγούμενο αυτός να παγώσει κατά κάποιο τρόπο να μην είμαστε φιλόδοξοι αλλά θα πρέπει να μην ξεχνούμε την καταβολή της μενούς διάκρισης, την ε, προώθηση της ισότητας. Αλλιώς κινδυνεύουμε να υπονομεύσουμε βασικό άξονα δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτές οι αρχές να μην ξεχνιούνται. Ισότητα και καταπολέμηση της δημιουργικής διάκρισης. Είπαμε δεν υπάρχουν πολλά χρήματα για νέες πρωτοβουλίες και άρα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τα κεκτημένα του ΣΥΠΗΝ να συνεχίσουν να τρέχουν αυτά τα οποία έχουν εγκριθεί, όπως με το πρόγραμμα Δάφνη, εδώ και κάποια χρόνια ε, ασχολούμεθα με αυτό και θυμάμαι επανειλημμένα σε πολλές ζητές για τον προπολογισμό ότι υπέστη επίθεση το πρόγραμμα Δάφνη. Άρα να εξασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσει να υπάρχει και θα βάλουμε φραγμό σε οποιαδήποτε προσπάθεια υπονομευσή του γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι τώρα σε τέτοιου καιρού κρίση, οι πιο ευάλωτε ομάδε του πληθυσμού να μην τους, παραμελούμε γιατί αυτοί χτυπιούνται από την κρίση περισσότερο. Άρα, να μην νύψουμε τα σχήρα μας και να πούμε «Απ, περικοπές λόγω της κρίσης, άστος αυτούς» γιατί αυτοί είναι οι πιο ευάλωτοι. Και οι γυναίκες πάντοτε είναι οι πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Επομένως, θα πρέπει να μελετήσουμε πώς έχουν επηρεαστεί από την κρίση οι γυναίκες και να δούμε πέρα από την κρίση πώς θα διεκπαιρεωθεί το θέμα του προϋπολογισμού γιατί εδώ και κάποιο καιρό η κρίση σοβεί, αλλά λίγα σκαρφιζόμαστε για το πώς θα την τερματίσουμε. Και έχουμε επίσης και διάφορες χώρες που εδώ είναι το πρόγραμμα, αλλά όπως η Σουδία και η Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχουν το ευρώ. Άρα πρέπει να δούμε πώς θα προστατεύσουμε αυτούς τους ευάλωτους της κοινωνίας. Και μην ξεχνούμε τη στρατηγική για το 2020, ανάπτυξη, θέση απασχόληση κλπ. Διότι εγώ θεωρώ και το ίδιο και η ομάδα των σοσιαλιστών ότι χρειάζεται η ανάπτυξη. Δεν χρειάζεται μόνο λιτότητα, άρα θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο όσον αφορά την απασχόληση των γυναικών. Πώς οι γυναίκες λοιπόν, πώς γυναίκες έχουν στο 62% σύμφωνα 75% ενεργείας των ανδρών και ότι σε μέσο όρο είμαστε ότι οι γυναίκες είναι, παίρνουν 16,4% από ότι οι άντρες για κάθε ώρα εργάσιμη επομένως Χρειάζεται όλο και περισσότερε γυναίκε να μπουν στην αγορά εργασία. Εάν θέλουμε το 75% που, έχουμε, που θέλουμε μέχρι το 2020 να το πετύχουμε σαν ε, ε, ρυθμό απασχόληση. Ιδάλω δεν θα βοηθήσουμε την οικονομία, ιδάλω δεν θα βοηθούν οι γυναίκε ε, από τα επιδόματα ανεργία. Άρα αυτό το οποίο χρειάζεται είναι αυτού του είδους τα τα επιχειρήματα να τα λάβουμε υπόψη, γιατί θα πρέπει έτσι να λάβουμε υπόψη αυτά τα επιχειρήματα που κατατείνουν στο πώς θα βοηθήσουν την οικονομία οι γυναίκες. Έχουμε επομένω όλα αυτά τα πιλωτικά προγράμματα και άρα θα έπρεπε με τη βοήθεια του κυρίου Λαβία να δούμε τι γίνεται με αυτά τα πιλωτικά προγράμματα, τι γίνεται με τις μονογονικές οικογένειες που είναι προηγουμένως κυρίως μονογονικές οικογένειες αποτελούνται από γυναίκες, πώς θα δουλεύουν, όλοι και περισσότερες είναι οι γυναίκες στην άλλη του φάσματος, γιατί βεβαίω θα πρέπει να δουλεύουν οι αλλά θα πρέπει και να συνεχίσουμε να δούμε και πώς ε, ανελίσσονται στη σταδιοδρομία τους και πώς αξιοποιούνται όλες τις δυνατότητές τους. Άρα, μην το ξεχνούμε αυτό. Παρά το ότι κινούμεθα μέσα σε αυτή την συγκυρία της κρίσης. Επίσης, πώ εκπροσωπούνται οι γυναίκε, πώ παρουσιάζονται οι γυναίκε από τα μέσα ενημέρωση, τι οικονομικέ συνέπειες έχει αυτό, τι γίνεται με τη βία ε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρόκειται για πρόγραμμα, project το οποίο δεν κοστίζει πολύ. Άρα αξίζει να το δούμε αυτό και να αφήσουμε τις περικοπές και αυστηρότητα στην άκρη. Τα στερεότυπα επίσης να τα καταρρύψουμε σε σχέση με το πρόβλημα της βίας και τέτοια πιλωτικά προγράμματα θέλω να υπάρξουν όμως θα έπρεπε να κάνουμε και άλλες προσπάθειες. Τη συμμετοχή στον πολιτικό βίο των γυναικών είναι η δουλειά μας, γιατί είμαστε Επιτροπή Ζητημάτων των Γυναικών. Άρα να δούμε τα θέματα της συμμετοχής, τα θέματα της παιδείας, εκπαίδευσης, τα ποσοστά αναλφαβητισμού και αυτό έχει οικονομικές ε, συνέπειες. τι άλλα τι άλλο θα μπορούμε να το, το, το τελεμπόριο βάρο γυναικών σε μέσω τρίτων χωρών, σε τρίτες χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πάντα με προβλημάτισε και το Λονδίνο είναι σταυροδρόμι αυτού του δουλεμπορίου ει βάρο των γυναικών. Όλα αυτά βεβαίω και σχετικά με τον προπολογισμό. Και μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα. χωρί αυτό να κοστίζει πολλά χρήματα. Είναι σημαντικό Θα σα δείξω τον αγώνα μας υπέρ των γυναικών και κατά την δυσμενών διακρίσεων τη βάρος του. Ευχαριστώ. Ο κύριο Λαβία ακόμη δεν ε, έφτασε. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα δύο λεπτών. Να επανέλθουμε πολύ γρήγορα. Επομένω μην κουνηθείτε παρακαλώ. Okay, we will uh, now start the meeting again. Να ξεκινήσουμε και πάλι με τη συνεδρίασή μας. Και λείπαμε που έπρεπε να τοποθετηθείτε πριν από τον ε, κύριο Λαβία. Βέβαια θέλαμε να εξοικονομήσουμε κάτι χρόνο, αλλά φυσικά αν το επιθυμείτε Μπορείτε να ξαναπάρετε το λόγο με την τοποθέτηση του κυρίου Λαβία. Είχατε την ευκαιρία να πείτε κάτι δύο φορές, έτσι λοιπόν αυτό είναι εξαιρετικό. Να σας καλωσορίσω κύριε Λαβία, έχετε το λόγο. Όπως ακούσατε, μόλις ξεκινήσαμε με το θέμα αυτό. Ακούσαμε την κυρία Χάνιμπολ, αλλά τώρα εσείς έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που είχαμε κάποια απόκληση στο χρόνο, αλλά εγώ είχα ενημερωθεί ότι έπρεπε να είμαι εδώ παρατέταρτο. Δεν καταρθέσαμε λοιπόν να συντονιστούμε πολύ καλά με το χρόνο. Όπως ξέρετε, η διαδικασία της έγκρισης του προπολογισμού για το 2013 ξεκίνησε στο Στρασβούργο με την έγκριση των κατευθυντηρίων γραμμών, το πρώτο επίσημο έγγραφο, ε, και πριν από την παρουσίαση του σχεδίου προπολογισμού από την Κομισιόν που θα γίνει μεθαύριο. Έτσι λοιπόν στις 25 του μήνα η Κομισιόν θα μας παρουσιάσει την πρόταση προπολογισμού του για το 2013. Είναι σαφέ ότι η έλευση μου σε αυτή την επιτροπή, όπως και το πέρασμα μου και από τι άλλε ε, επιτροπές, ε, ε, έκανε μία απευθεία σύνδεση με όλες τις επιτροπές που φυσικά θεωρούν την διαδικασία των μεμονωμένων τομέων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και έχουν πολύ περισσότερη αρμοδιότητα από όσο θα μπορούσε να έχει η Επιτροπή Προπολογισμού, η οποία αντίθετα βλέπει το θέμα συνολικά. Έτσι λοιπόν η παρουσία μου εδώ θέλει να ε, δημιουργήσει μια ισχυρή σχέση με όλες τις επιτροπές για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε όλοι μαζί και να καταλήξουμε στο τελευταίο προπολογισμό του επταετούς προγράμματος. Ε, όλοι ε, θα γνωρίζετε ότι θα υπάρχουν αρκετές δυσκολίες για την έγκριση αυτού του προπολογισμού και γιατί γιατί αν ε, αφενός ε, ζούμε σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, έχουμε μια διαδεδομένη κρίση, έχουμε μια κατάσταση όπου τα κράτη-μέλη σε εσωτερικό επίπεδο αντιμετωπίζουν μια σειρά δυσκολιών και αφετέρου σε κοινοτικό επίπεδο, ε, στο πλαίσιο της πολιετούς χρηματοδότησης πρέπει να ολοκληρώσουμε πολλά προγράμματα. Και καθώς τα προηγούμενα χρόνια είχαμε πολύ περισσότερες ε, αναλήψεις υποχρεώσεων ε, παρά υποχρεώσεις πληρωμένων. Τώρα ε, βρισκόμαστε σε μια διαφορετική κατάσταση. Έτσι λοιπόν, ολόκληρο το σύστημα Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένα δεν θα μπορεί παρά να παρουσιάσει μεθαύριο ένα πρόγραμμα προϋπολογισμού, ένα προσχέδιο προϋπολογισμού που θα χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις αναγκαιότητες ε, κονδυλίων για πληρωμές και όλοι θα γνωρίζουν ότι πέρσι και προσπαθώ τώρα να ενημερώσω όλους τους συναδέλφους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε πάρα πολλές δυσκολίες στην υλοποίηση των πληρωμών σκεφτείτε ότι το τελευταίο μήνα είχαμε ε, κάποιες δεσμεύσεις κεφαλαίων για το 1α για την έρευνα, για το 1β για 16 δισεκατομμύρια ευρώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν σε θέση με ε, του πόρους ε, που είχε στον προπολογισμό να καταβάλει μόνο 5 δι. Αυτό σημαίνει ότι 11 δι πληρωμών που θα έπρεπε να γίνουν στα πλαίσια του οικονομικού έτου 2011 με τον προπολογισμό του 2011 μεταφέρθηκαν στο 2012. Έτσι λοιπόν ήδη στον προπολογισμό του 2012 ξεκινήσαμε μία έλλειψη κονδυλίων για πληρωμέ και υπάρχει κίνδυνος να υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα και να έχουμε και άλλη μεταφορά κονδυλίων για το 2013. Έτσι λοιπόν ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι ιδιαίτερα ρεαλιστική ε, και να ε, ε, μην ε, ε, αναφερθεί στον τύπο μια σειρά εκπόνηση κονδυλίων για την περίοδο κρίσης, γιατί φυσικά δεν έχουμε τη δυνατότητα να κλείσουμε το προπολογισμό και με τις κατευθυντήριες γραμμές ζητήσαμε στον επόμενο προπολογισμό να έχουμε ένα προπολογισμό που θα κατευθύνεται προς την ανάπτυξη και την απασχόληση και προς τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Γιατί έχουμε, αυτά είναι τα δύο στοιχεία που έχουμε και θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Και βέβαια έχουμε και μία σειρά άλλων ε, θεμάτων που πρέπει εμείς από κοινού πρέπει να καθορίσουμε ως προτεραιότητες. Γιατί αυτές είναι μεγάλες ε, προτεραιότητες για το μέλλον προϋπολογισμού... αλλά εμείς πρέπει να δούμε τι θα γίνει σε κάθε γραμμή προπολογισμού. Και έτσι θα αρχίσουμε από σήμερα να εργαζόμαστε όλοι από κοινού για να ε, προκαθορίσουμε την εντολή για τον τριμερή διάλογο. Και φυσικά είμαι εδώ για να σας να συμμετάσχετε σε αυτή τη διαδικασία, για να σας ζητήσω, να σας ρωτήσω ποιες είναι οι προτεραιότητες που θέλει να παρουσιάσει η δική σας επιτροπή και να υπογραμμίσω ότι σε μία περίοδο κρίσης θα πρέπει να είναι υπεύθυνο ο προπολογισμό μας, όπως και τα αιτήματά μας ως κοινοβούλιο. Δεν ε, μπορούμε να σκεφτόμαστε να ζητάμε περισσότερα σε κάποιες γραμμές προπολογισμού αν δεν μπορούμε να εντοπίσουμε και κάποιες αρνητικές προτεραιότητες. Γιατί αν είναι αλήθεια και όπως είναι αλήθεια ότι ορισμένα ε, προγράμματα θα ενισχυθούν από την άλλη ε, πρέπει να είμαστε και ικανοί να προσδιορίσουμε αν υπάρχουν προγράμματα που δεν έχουν τόσο καλές επιδόσεις, που είναι λιγότερο αποτελεσματικά και να προτείνουμε κάποιες μειώσεις. Έτσι λοιπόν, για να συμμετέχουν όλοι, θα συναντήσω όλους τους ειδικού ε, εισηγητές, δηλαδή όλους τους εισηγητές που έχουν αναλάβει ε, το συγκεκριμένο θέμα στις 9 Μαΐου, προκειμένου να συλλέξω από όλους όλες τις ενδείξεις και τις πληροφορίες και ε, να μπορέσω να συμπεριλάβω τα σχολιά τους στην εντολή για τον τριμερή διάλογο και να ε, τους επικαιροποιήσω και για την πορεία των εργασιών. Και επίσης θα μιλήσουμε και για τις προσκευαστικές δράσεις και τα πιλωτικά προγράμματα, αλλά μου φαίνεται ορθό ήδη από το στάδιο αυτό να σας πω ποια είναι η διαδρομή που θα ακολουθήσουμε. Γιατί σε μια περίοδο κρίσης ε, όπου έχουμε περιορισμένους πόρους δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε αυτού μα να μπλοκάρουμε πόρους για ε, project που στη συνέχεια δεν θα εφαρμοστούν. Έτσι, να δεσμεύσουμε πόρου δηλαδή για σχέδια που δεν εφαρμοστούν. Έτσι λοιπόν, καταρχήν, θα υποβάλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι αρχέ Ιουνίου ένα κατάλογο με πιλωτικά ε, σχέδια που θα θέλει να παρουσιάσει κάθε επιτροπή προκειμένου να υπάρξει μια προκαταρκτική αξιολόγηση από την πλευρά της Κομισιόν. Γιατί η προκαταρκτική αξιολόγηση, γιατί αν ένα πιλωτικό σχέδιο δεν εφαρμοστεί σύμφωνα με την Κομισιόν, ε, γιατί ήδη υπάρχει μια γραμμή προπολογισμού που καλύπτει αυτό το είδος της δραστηριότητας και έτσι λοιπόν δεν θα μπορεί να αναπτυχθεί και δεν θα πρέπει να δεσμεύσουμε πόρους του προπολογισμού για αυτή τη συγκεκριμένη project, για τη συγκεκριμένη γραμμή δραστηριότητα και ε, τελικά δεν εφαρμοστεί το πρόγραμμα, τότε δεσμεύουμε του πόρου, ενώ θα μπορούσαμε να του έχουμε χρησιμοποιήσει κάπου αλλού. Έτσι λοιπόν, αν από την αρχή, ε, αν σας ζητήσουμε να υποβάλλετε τα πιλωτικά σχέδια και θα έχουμε μια προθεσμία στα τέλη Μαΐου, έτσι ώστε στις αρχέ Ιουνίου η Επιτροπή Προπολογισμού ε, που συλλέγει όλα τα project ε, να μπορεί να τα στείλει στην Εκτελεστική Επιτροπή να μπορέσουμε έτσι μέσα στον Ιούλιο να δούμε αν είναι εφικτό να υλοποιηθούν ε, αυτά τα project και θα έχουμε τα γράμματα ε, D, C, B και A. Τα D θα είναι αυτά που δεν μπορούν να εφαρμοστούν γιατί έχουμε ήδη μία γραμμή υπολογισμού. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που καλύπτει αυτή τη δραστηριότητα. Έτσι λοιπόν χάνεται η φύση του πιλωτικού σχεδίου γιατί αυτό ήδη υλοποιείται. Τώρα, τα CBKE project θα είναι τα εξή. Τα C θα χρήζουν βελτιώσεων, ε, τα B κάτι λιγότερο, ενώ τα A, τα Α ε, βρίσκουν όλου σύμφωνους ε, και μπορούν να εφαρμοστούν. Κατόπιν λοιπόν της αξιολόγησης της Επιτροπής θα μπορέσουμε να τα τροποποιήσουμε και να τις συμπεριλάβουμε έτσι ώστε να έχουμε προγράμματα που θα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν και αυτά θα αποτελούν μέρος του συνολικού πακέτου που θα εγκρίνουμε όταν θα συζητήσουμε την τελική έγκριση του προπολογισμού. Έτσι λοιπόν, εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο, πέρα από το θέμα της προθεσμίας. Νομίζω ότι βέβαια ως γραμματεία έχετε ενημερώσει. Έχουμε την 25η Απριλίου την παρουσίαση του σχέδιου προπολογισμού από την ε, Κομισιόν 9 Μαΐου, συναντήση με τους ειδικούς συζητητές ε, στις αρχές Ιουνίου, παρουσίαση ε, των πιλωτικών σχεδίων και στη Σύνοδο του Ηλίου ψηφοφορία για την αντολή για το διάλογο, τον τριμερή διάλογο και πιθανότατα την πρώτη-δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου θα έχουμε μια προθεσμία για την παρουσίαση των τροπολογιών. Και στη Σύνοδο του Οκτωβρίου θα πρέπει να ψηφίσουμε τη θέση μας ε, ε, στον προπολογισμό και κατόπιν έχουμε 21 μέρες για την συνδιαλλαγή, για την ε, συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Αυτή είναι η διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθήσουμε αν όλα πάνε καλά, τότε θα έχουμε την έγκριση του προπολογισμού. Σας ευχαριστώ. Ja, det är den som lever får veta det. Ο πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα, περιμένουμε και να δούμε τι θα γίνει. Και τώρα ξαναδώσουμε τη σκητάλη τη κυρία Χανιβόλη, αν βεβαίω θέλει, να συμπληρώσει αυτό το οποίο είπε προηγουμένω. Βέβαια να μην επαναλάβει τα ίδια, αλλά ίσω ίσως δεν ασχολεί αυτά τα οποία ακούσαμε από εσά. Ναι, ναι, πρόεδρε, σα ευχαριστώ. Δεν ε, Ακούσατε τι είπα προηγουμένω, αλλά να δούμε, να σας αναφέρω τώρα τι θα ήθελα να περιλάβετε στο κείμενο. Ε, γιατί ένας από τους βασικούς τομέας που θέλουμε ότι θα πρέπει να είναι προτεραιότητα είναι η απασχόληση των γυναικών. Ε, κάτι το οποίο βεβαίως ε, τις κάνει απολύτω των ανδρών και άρα έχουμε ε, τη 2020 βεβαίως Έχουμε και την ε, ανεργία των νέων, αλλά αν δεν καλύψουν και τις γυναίκες, οπότε θα ήθελα ε, αυτό να το πείτε σε οτιδήποτε πρότεινε για τον προπολογισμό και νομίζω ότι αυτό γενικά θα είναι θετικό. Άρα φαντάζομαι ότι γίνεται. Κάτι το οποίο, δεν είπαμε προηγουμένω είναι το, το, το, το, το θα έχουμε mainstreaming ένταξη στι όλε τι πολιτικέ, ε, τα θέματα των δύο φύλων, τη ισότητα σε όλες τις δράσεις της Ένωσης. Και να μην το συζητάμε μόνο εμείς εδώ σε αυτήν την Επιτροπή για τη θέση των γυναικών να γίνει ευρύτερα πολιτική της Ένωσης. Έτσι να τα βλέπουν όλες οι Ένωσες τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι αυτό θα φέρνει τον πρωτοβουλίο, επομένω παρακαλώ να το συμπεριλάβετε τώρα. Κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε όταν μιλούμε για τις όλες αυτές τις ομάδες, σας είπα και προηγουμένω, ότι από τη βάση της εμπειρίας με την Επιτροπή, στην οποία δουλεύω εδώ για 10 χρόνια πάρα πολύ συχνά, το πρόγραμμα Δάφνη έχει θεωρηθεί ε, κάτι το οποίο μπορεί να επιδέχεται περικοπές. Δεν είναι όμως αλήθεια αυτό, διότι πρόκειται για πάρα πολύ σημαντικό ρόλο τον οποίο επιτελεί. Όχι, δεν θέλουμε βία κατά ουδενός και φυσικά όχι κατά των γυναικών και το πρόγραμμα Δάφνη είναι πολύτιμο σε σχέση με το πώς θα βάλουμε να φραγμό σε αυτή τη βία. Επομένως παρακαλώ να σταματήσουν αυτές οι απόπειρες υπονόμευσης, να μην ε, τις ξαναδούμε. Επομένως, τώρα να δούμε και άλλες ευάλωτες ομάδες όπως οι μονοφανικές οικογένειες να βοηθηθούν. να τους φροντίσουμε με πολλές Τι Ποιες προσκευαστικές δράσεις να δούμε. Πώς, πώς, πώς θα συμπεριληφθούν και αυτές οι μονογονικές οικογένειες. Τι γίνεται επίση αν ε, έχουν ανώτερες και ανώτατε θέσει στο προσωπικό των εταιρεών οι γυναίκε, Θέλουμε να συμμετέχουν περισσότερο οι γυναίκες σε αυτό το επίπεδο διοίκηση των εταιρεών. πώς προβάλλονται οι γυναίκες ε, στα ΜΜΕ, πώς τις διαφημίσεις, γιατί υπάρχει σχέση μεταξύ αυτής της εικόνα τη γυναίκας και της άρχης βίας βάρος της. Και αυτό όλη την Ευρώπη και υπάρχουν επίσης και στερεότυπα. Μην ξεχνάμε τι, υπόψη, τι έχουν υποστεί οι γυναίκες, τι έχουν περάσει. Λοιπόν αυτά σε αδρές γραμμές για το τι θέλουμε να αναπτύξετε. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να σέβεστε, να προωθείτε την αξία αυτή στην Ευρωπαϊκή για τα καταπολέμηση δηλαδή, της διμηνής διάκρισης. Να μην ξεχνούμε καθόλου αυτό, αυτό το, αυτή, τον αγώνα μας, ακόμα και σε εποχές κρίσης. Tack, eh, tack för det och då går ordet till fru Matera, varsågod. Grazie, Presidente. Κυρία Ματέρα, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το συνάδελφο τον κύριο Λαβία που παρευρίσκεται εδώ σήμερα και που υιοθέτησε την αρχή της ε, υπευθυνότητας και της διαφάνειας καθώς μπλέκει στη διαδικασία του προπολογισμού όλες τις επιτροπές και τους εισηγητές των Μονομένων Επιτροπών. Εγώ μιλώ όχι μόνο ως αντιπρόεδρος αυτής της επιτροπής αλλά και ως κοιόδης ε, της ομάδας του ΕΛΚ σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό αυτής της επιτροπής όλοι μας εκτιμήσαμε το γεγονό ότι φέτο μεταξύ των κατευθυντηρίων γραμμών ε, που παρουσιάστηκαν πριν από λίγου ε, μήνε, επικεντρωνόμαστε φέτο στον προπολογισμό του 2013 στου νέου και στο τι μπορεί να γίνει για την απασχόληση των νέων και κυρίως ε, στην υποστήριξη στις μικρές και μεσές επιχειρήσεις, καθώς ε, το 2002 στο 2010 το 80% των νέων θέσεων εργασία ε, δημιουργήθηκε στις μικρές και μεσές επιχειρήσεις και επίσης στην υποστήριξη της κινητικότητας. Η κινητικότητα έχει να κάνει με την υποστήριξη των τομέων της κοινοτομίας και της έρευνας που μπορεί να ανοίξει νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Έτσι λοιπόν, ε, ω σκιώδη ε, για την Επιτροπή αυτή, για το θέμα του προπολογισμού, έχω την ε, ευκαιρία να συζητώ με τον κύριο Λαβία και να μπορώ να υπογραμμίσω κάποιε από τι πτυχέ που κατά τη γνώμη μου λείπουν από αυτό το σχέδιο προπολογισμού. Καταρχήν, η πιο κατάλληλη χρηματοδότηση για το θέμα της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων για την περίοδο 2010-2015 και οθέτηση ενός προϋπολογισμού για την ισότητα των δύο φύλων για να προωθήσουμε καλύτερα το θέμα της ισότητας και επίσης ιδιαίτερη προσοχή στις γραμμές προϋπολογισμού 2013 και στον αριθμό των ε, ευάλωτων γυναικών που ένα και αυξάνονται δηλαδή με αναπηρία, τις μετανάστριες, γυναίκες που ενήκουν σε εθνοτικές μειονότητες και σε μόνες γυναίκες και στις μόνες μητέρες. Είμαι ικανοποιημένος που η συνάδελφος Χάνιμπολ μίλησε για αυτή την κατηγορία. Και τέλος, ε, είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε το πρόγραμμα Δάφνη ε, για να εγγυθούμε όλα τα μέτρα για την καταπολέμηση της ε, βίας κατά των πιο δύναμων, κατά των γυναικών και το πρόγραμμα Progress για την προώθηση της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Σε όλα αυτά όπως ε, σωστά υπογράμμισες πριν, σε ευχαριστούμε που μας έχεις δώσει καλές ενδείξεις ε, για να μπορέσουμε να πράξουμε έτσι τουλάχιστον φέτος ε, ένα πιλωτικό σχέδιο αν και θα θέλαμε κάτι περισσότερο, να μπορούσε να γίνει αποδεκτό. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι θα τα δεκτούν ευχαρίστω όλοι οι συνάδελφοι όλα αυτά. Μα αναφέρετε και αυτή είναι η κύρια ε, επιθυμία που έχουμε εμεί ω Επιτροπή ΦΕΜ των δικαιωμάτων των γυναικών και σε ευχαριστούμε για το μεγάλο κουράγιο που έδειξες και για τον τρόπο που ε, αντιμετώπισες αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Ευχαριστώ Τζοβάνι και ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ δώσω στον κύριο Λαβία το λόγο για να ολοκληρώσει. Θα ήθελα να πω δύο λόγια κι εγώ. Συστούμε τον προπολογισμό, τη δημοσιονομική κρίση. Βλέπουμε ότι είναι δύσκολο να εξασφαλίσουμε πόρους και κυρίως σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την ε, ε, ισότιμη μεταχείριση, με την καταπολέμηση των διακρίσεων. Όλα αυτά βλέπουμε ότι ξεπερνούν το 12 του προϋπολογισμού. Είναι μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην εξέλιξη, στην ανάπτυξη ανθρωπότητας και έτσι έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία κοινωνική αλλά και οικονομική. Από την άλλη θα μπορούσαμε να συστήσουμε και τις πιο βραχυπρόθεσμες ε, προοπτικές. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία ε, κοστίζουν πολλά. Και εάν ε, σκεφτούμε καθαρά οικονομικά, με ορσόρους οικονομικούς, δηλαδή αγνοώντας την κοινωνική διάσταση, θα παραγνωρίσουμε πολλές πτυχές του προβλήματος. Δεν θα μπορέσουμε να ε, τιμήσουμε πολλές από τις πτυχές του προβλήματος. Αυτό ήθελα να δώσω εγώ σαν παρατήρηση από πλευρά μου, αλλά βέβαια έχετε το λόγο κύριε Λαβία για να ολοκληρώσετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και για αυτά τα τελικά σχόλια που κάνατε και πραγματικά τα όσα προγραμματίζεται μας καλούν να παρουσιάσουμε έναν υπεύθυνο προπολογισμό λαμβάνοντα υπόψη και την πτυχή του φίλου σε μια περίοδο κρίσης ενώπιον όλων. Τελικά ε, σήμερα ε, τα κράτη-μέλη δίνουν πολύ μεγάλη προσοχή στη συγκράτηση των δαπανών, γιατί τα 27 κράτη-μέλη ε, όλα κάνουν εσωτερικές θυσίες, ε, πολύ μεγάλες θυσίες στο εσωτερικό επίπεδο και έχουν δυσκολία ώστε να συνεισφέρουν περισσότερο στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό πρέπει να μας οθήσει στο να υλοποιήσουμε έναν υπεύθυνο προπολογισμό Ευρωπαϊκής Ένωσης, έναν σωστό προπολογισμό και να μπορεί να χρησιμοποιούνται στον εδόν καλύτερο υπόρρο που διαθέτουμε. Είναι σαφές ότι εντός και μεταξύ των προτεραιοτήτων των κατευθυντηριών γραμμών θέλαμε να αναφέρουμε μόνο γενικές προτεραιότητες. Τώρα στην εντολή του τριμερούς διαλόγου φυσικά θα μπούμε στις λεπτομέρειες και θα ε, αναφέρουμε τις προτεραιότητες ε, με ιεραρχική σειρά. Εγώ σας ευχαριστώ για τις ενδείξεις που μου δώσατε από την πρώτη ανταλλαγή απόψεων και σημειώνω κάποια πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Συντητούτο για την Ισότητα των Διοφύλων, σε σχέση με τη δυνατότητα της χρήσης και των διαθροτικών ταμείων για την προώθηση των πολιτικών που αφορούν την ισότητα των διοφύλων και ε, τα περισσότερα ζητήθηκαν σε σχέση με το πρόγραμμα Δάφνη για ορισμένε πτυχέ και το πρόγραμμα Progress για άλλε πτυχέ και υποστήριξη και κάποιων πολιτικών. που έχουν να κάνουν με τη συνεργασία για την ανάπτυξη σε σχέση με ορισμένα μέτρα που λαμβάνονται στις τρίτες χώρες ε, κατά παραδείγματος χάρη του ακριτηρισμού των γεννητικών οργανών των γυναικών και τη ε, καταπολέμησης τη εμπορία ανθρώπων. Είναι σαφέ ότι υπάρχουν μία σειρά προτεραιότητε που έρχονται από τη δική σα Επιτροπή όπως ε, το να υπάρχει και μία σειρά ε, σχεδίων πιλωτικών που να αφορούν και την ισότητα των δύο φύλων. Όμως ε, εμείς ε, δεν μπορούμε να δεσμεύσουμε πόρους για πρωτοβουλίες που δεν θα αναπτυχθούν στη συνέχεια, οπότε πρέπει να το εξετάσουμε και αυτό. Σας ευχαριστώ για αυτές τις πρώτες προτάσεις, αυτή την πρώτη ενταλλαγή απόψεων και φυσικά από εσά αναμένουμε αυτές τις συγκεκριμένες προτάσεις ε, που θα αναφέρονται στη γνωμοδότηση που θα καταθέσετε στην Επιτροπή Προπολογισμών και φυσικά είμαστε στη διάθεσή σας να τις λάβουμε υπόψη και στην εντολή για τον τριμερή διάλογο και στην συνέχεια των διαπραγματεύσεων που θα μας οδηγήσουν στη συνέχεια του χρόνου στην έγκριση του προπολογισμού. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν για τις μελλοντικές σας συνεισφορές και φυσικά θα έχουμε και τη συνεδρίαση με τους συντονιστές από όλες τις ειδικές επιτροπές για να προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε υπεύθυνα τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θέλουμε να αναφέρουμε στην άλλη αρχή του προπολογισμού για την τελική συνδιαλλαγή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δώσετε να συζητήσουμε και βεβαίω εμείς θα κοιτάξουμε να δώσουμε μια απάντηση σωστή και σοβαρή. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα, για τις προθεσμίες κατάθεση τροπολογιών στη γνωμοδότηση της κυρίας Χάνιμπολ δεν έχουμε προσδιορίσει ακόμα ημέρα. Θα σας ενημερώσουμε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Τώρα κάνουμε μια μικρή διακοπή δύο λεπτό, για να επανέλθουμε με την κοινή συνεδρίαση. Okay. Um, good afternoon. Καλησπέρα σας. Ξεκινούμε τώρα τη συνεδρίαση. Και εγώ θα γυρίσω στην σουηδική γλώσσα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους προς την, ε, στην κοινή μας αυτή συνεδρίαση μεταξύ της Επιτροπής των Γυναικών και της Νομικής Επιτροπής. Με χαρά βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον και υποστήριξη για την προσπάθεια αυτή. Είναι πολύ σημαντική για την ε, Επιτροπή μας η συνεργασία και η δυνατότητα για μια κοινή πρόταση είναι σημαντική για τις γυναίκες και για την ισότητα των ευκαιριών εν γέννη. Ιδιαίτερα λοιπόν χαιρόμαστε για αυτή την ευκαιρία που προσφέρεται και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τις παρουσιάσεις. Η συγγετρία πρώτα παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι ιδιαίτερα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιμένω την συζήτηση των τροπολογιών. Εδώ έχουμε να κάνουμε την επέκταση του ε, πεδίου προστασίας ένα τομέα δηλαδή πολύ συγκεκριμένου, με πολύ συγκεκριμένα ωφέλη και πλεονεκτήματα για τον πολίτη, την πολίτη της Ευρώπης. Εφόσον βέβαια τον χειριστούμε σωστά τον χώρο αυτό, το πεδίο αυτό. Εδώ έχουμε να κάνουμε την προστασία του θύματος με τον ε, κανονισμό που έχει συζητηθεί στις διάφορες επιτροπές ήδη και τώρα προχωρούμε λίγο πολύ στην πτυχή την αστική, του αστικού δικαίου, τον κανονισμό δηλαδή για την αμοιβαία αναγνώριση των μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις. Πολλά πράγματα πιστεύω θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε, να κερδίσουμε για τα θύματα εάν μπορούσαν ε, να κυκλοφορούν στο βαθμό του δυνατού ελεύθερα στην Ευρώπη. Γι' αυτό όμω χρειάζονται και συγκεκριμένα μέτρα και γι' αυτό χαιρόμαστε ιδιαίτερω για τη συνεργασία μεταξύ Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων και Επιτροπή των Γυναικών, διότι οι μεν γνωρίζουν καλά τα μέσα που είναι διαθέσιμα, η δε όμως, η δε επιτροπή γνωρίζει πολύ καλά τα ζητήματα, την ουσία του προβλήματος. Τα θέματα που θα να επιλύσουμε. Και ελπίζουμε ότι θα λειτουργήσει καλά αυτή η συνεργασία για να διατυπώσουμε με τρόπο ευφύ και αποτελεσματικό το νομοθέτημα αυτό. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σταματήσω την ε, παρέμβασή μου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρος. Και τώρα να δώσουμε στους συζητητές τον ε, λόγο. Πρώτα πρώτα κυρία Παρβάνοβα, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ να σας αναφέρω ότι είναι πάρα πολύ στενή η συνεργασία μας. Προσωπεί την Νομική Επιτροπή ο κύριος Λόπες. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να παραστεί. Πάντως όλα όσα θα σας πω τα ασπάζεται εκείνος και οι συνεργάτες του. Και είναι χρήσιμη αυτή η συνεργασία. Γιατί έτσι συμβάλλουν στη διαμόρφωση τη αρχική πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε και έτσι ευθυγραμμιζόμαστε με όλα όσα πρεσβεύουν όλοι οι συνάδελφοι και στι δύο επιτροπέ. 40 είναι συνολικά οι τροπολογίε που υπευλήθησαν. Οι περισσότερε από αυτέ είναι στο δίμηκο σχήματο με το σχέδιο κειμένου μα. Και επίση έτσι βέβαια αυτό υποστηρίζει υποστηρίζει, προωθεί την έκθεση και μπορούμε και εμείς να δουλέψουμε καλύτερα τις τροπολογίες και να βελτιώσουμε την πρόταση της Επιτροπής. Τώρα, το ανακτήριο λάκτισμα. Για να δούμε. Ποια είναι τα σημεία στο οποίο επικεντρώνονται περισσότεροι συνάδελφοι. Να τονίσουμε. Ότι αυτά όλα έχουν σχέση με κάποια μέσα προστασίας. Και να σας πω τις τέσσερις ομάδες τροπολογιών που έχουμε σε σχέση με το σχέδιο κειμένου. Πρώτα πρώτα. Απλούστευση της διαταγής αναγνώρισης. Η διαδικασία αναγνώρισης και η χρήση των πιστοποιητικών. Στο 72 λέει για κάποιους σαφείς στόχους. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μεγαλύτερη προστασία για τα θύματα. Να είναι πιο απλή η ε, διαδικασία προστασίας για τα θύματα. Παντού. Αυτόματο σύστημα διαβίβασης για το πιστοτικό προστασίας. Και όταν ο προστατευόμενος δεν βρίσκεται στην χώρα προέλευσης να μπορεί να υποβάλει αίτηση με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικά ή άλλο, για να του χωρίζει το πιστοποιητικό και έτσι καλύπτουμε όλες τις δυνατότητες για να γίνει ευκολότερη η όλη διαδικασία. Επίσης, μέσω του εθνικού δικαίου, σε κηδεμόνα, έχονται την επιμέλεια, εκπρόσωπο να διαβάζεται αυτό. Το 63 επίση. Και αυτό ευθυγραμμίζεται με τι δικέ μα προτάσει. Και λέει για μια βάση δεδομένων σε την Ευρωπαϊκή Ένωση, κοινή. Έτσι, οι, ευρωπαϊκέ οι εθνικές αρχές θα έχουν πρόσβαση εύκολη σε αυτή τη βάση δεδομένων. Θα έχουν αποτελεσματική προστασία. Διασυνοριακή επίση, δεύτερη ομάδα τα δείγματα, τα, συγγνώμη, τα θύματα της βίας μεταξύ των δύο φίλων. Ευχαριστούμε για τις τροπολογίες, γιατί λέει για τα θύματα αυτής της βίας. Και μετά έχουμε την τροπολογία 87, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται εδώ με αυτές τις διατάξεις που ζητούν για την ευθυγράμμιση των προτύπων, των στάνταρ τέλο πάντων, προστασίας για τα θύματα της βίας μεταξύ των δύο φύλων. Έχουμε την οδηγία που βρίσκεται στη φάση του τριμερού διαλόγου και προσπαθούμε να ευθυγραμμίσουμε, να συντονίσουμε με την οδηγία και αυτές τις τροπολογίες με αυτό το κείμενο. Επίσης συμφωνούμε και με τις ε, προτάσεις που λένε για εξειδικευμένη κατάρτιση των ε, κρατικών υπαλλήλων σε σχέση με τα πρόσωπα που, των οποίων κινδυνεύει η σωματική ψυχολογική ακυρότητα, όπως λέει το 86. Επίσης, λέμε εδώ τις οργανώσεις, την κοινωνία των πολιτών, κάποιες θελοντικές οργανώσεις, όλοι αυτοί που έχουν συμβάλει και έχουν διευκολύνει τη ζωή των θυματών σε σχέση με τη γραφειοκρατία ή σε σχέση με το να ε, αναλαμβάνει ξεχωριστά η κάθε διοίκηση να σε αυτές τις υπηρεσίες θα πρέπει σε σχέση με μετάφραση και διερμηνία. Εκείνοι που δεν μιλούν τη γλώσσα της διαδικασίας όσον αφορά την αναγνώριση να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μετάφραση και διερμηνία. Και επίσης αυτό να αφορά ότι άλλα έγγραφα τους κοινοποιούνται. Αυτό είναι η τροπολογία 64. Τελευταία ομάδα συνειδητοποίηση, ενημέρωση, ούτως ώστε όλοι να έχουν τα δικαιώματά τους και επίσης να υπάρχει η ανεμπόδιστη παροχή της προστασίας και να υπάρχει μια τέτοια καμπάνια ενημέρωσης, όπως λέει η τροπολογία 86. Τέλος, θετικές οι διατάξεις που αφορούν την συλλογή δεδομένων. Ιδίως όπου Ε, μας απασχόλησε αυτό στο πρώτο τμήμα εκείνες τις μελέτες που είχαμε εξετάσει για την βία μεταξύ των δύο φύλων. Πώς δηλαδή θα πάρει συγκρισιμότητα μεταξύ των δεδομένων που συλλέγουν τα κράτη-μέλη. Να δούμε και τι ανάλυση θα γίνει για τις πληροφορίες της τροπολογίας 89 όσον αφορά το πώς λειτουργεί ο μηχανισμός αυτής, της, αυτού του πιστοποιητικού και πώς μπορεί να βελτιωθεί η διαδικασία. Ευχαριστούμε και περιμένουμε πώς και πώς τη δική σας συμβολή. Να βρούμε συμβαστικές τροπολογίες και να βελτιώσουμε την πρόταση της Κομισιόν. Tack så mycket för det och då ger jag ordet till eh, kommissionens representant fru Claudia Hahn. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Claudia Hahn, την εκπρόσωπο της Κομισιόν. Yes, thank you, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Κομισιόν ε, καταρχήν θέλει να ευχαριστήσει και τους δύο συγκεκριτές για την εξαιρετική συνεργασία. Είχαμε πάρα πολύ καλή επικοινωνία Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι με την έκθεση και με τις τροπολογίες που έχουμε επιτάπητος. Οδεύουν σαστός ε, προς ε, την επίτευξη του συνολικού στόχου της Κομισιόν ε, και ε, φυσικά, αν λάβουμε υπόψη και την οριζόντια οδηγία τα θύματα, θεωρούμε ότι για εμείς ως Κομισιόν συμφωνούμε με το Κοινοβούλιο στο στόχο να ενδυναμώσουμε τα δικαιώματα των θυμάτων σε αυτό το σημαντικό ζήτημα, σε αυτό το σημαντικό φάκελο. Δεν ε, μπορώ να σας πω πολλά για το τι συμβαίνει στο Συμβούλιο, αλλά στις διαπραγματεύσει του Συμβουλίου υπάρχουν κάποια τεχνικά ζητήματα που πρέπει να επιληθούν. Δεν έχουν επιληθεί όλα, δεν αντιμετωπίζονται όλα στις ε, τροπολογίες του Κοινοβουλίου. Υπάρχουν ορισμένα πολύπλοκα θέματα. Είναι πολύπλοκα επειδή οι δικαστικές σε ορισμένα κράτη-μέλη είναι αρμόδιες οι δικαστικές αρχές, ενώ σε άλλα κράτη-μέλη είναι η αστυνομία υπεύθυνη και έτσι αυτό θίγει την αμοιβή εμπιστοσύνη μεταξύ των αρχών αυτών και αυτό είναι κόκκινη γραμμή για την Κομισιόν και εμείς ε, πιστεύουμε ότι ε, θα πρέπει να τη σε εφαρμογή όλα τα μέτρα προστασίας για να έχουμε αποτελεσματική προστασία των θυμάτων. Θέλουμε να συμπεριλάβουμε όλα τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται και από τις δικαστικές αρχές ή από τις αστυνομικές αρχές ή από ένα δήμαρχο, παραδείγματο χάρη. Και υποστηρίζουμε ισχυρά οικονομικά δικαιώματα και ξέρουμε ότι συμφωνεί το Κοινοβούλιο με την ενίσχυση των δικονομικών ε, δικαιωμάτων. Υπάρχουν ορισμένα θέματα που έχουμε ήδη συζητήσει σε τεχνικό επίπεδο όπου όμως εξακολουθούμε να πρέπει να ελεγξούμε την δυνατότητα υλοποίηση ε, ορισμένων τροπολογιών. Έχουμε δύο θέματα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να αποφύγουμε ε, να έχουμε επικαλύψει με τη δουλειά που γίνεται στην Οδηγία προστασία των Θυμάτων και έχουμε κάποιες καλές προτάσεις επιτάπητος. Και για να είμαι απολύτω ειλικρινής, ε, εξακολουθούμε να έχουμε κάποια μικρή ανησυχία για τη νομική βάση δεν έχουμε λάβει την τελική καθοδήγηση από τη δική μας νομική υπηρεσία και καθώς αυτό είναι ένα εργαλείο αμοιβαίας αναγνώρισης, εξακολουθούμε να ε, ελέγχουμε αυτή τη στιγμή σε ποιο βαθμό μπορούμε εδώ να συμπεριλάβουμε όλες αυτές, αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες της υποστήριξης της μετάφρασης, Τη οργάνωση Υποστήριξη υποστήριξης των θυμάτων. Η Κομισιόν, να σα διαβεβαιώσω, 100% είναι υπέρ αυτών των ιδεών επί τη ουσία, αλλά εξακολουθούμε να περιμένουμε τη γνωμοδότηση τη νομική υπηρεσία μα για το αν είναι δυνατό, αν είναι εφικτό να υλοποιηθούν κάποιε από αυτέ τι τροπολογίε. Αλλά βάζουμε τα δυνατά μα για να ξεύρουμε μια καλή λύση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα θύματα. Ανυπομονώ λοιπόν για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις και είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι θα πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο ε, στους βουλευτές. Κύριε Παπαδοπούλου. Thank you very much. Ευχαριστώ. Από ό,τι κατανοώ, η Κομισιόν έχει την καλή βούληση συναισθητήσει πολλές από τι τροπολογίε μας, ε, επειδή, όπω είπαν ε, και τα συγκεκριτές, μέσω της ε, κυρίας Παραβάνουα, όλες οι τροπολογίε που παρουσιάστηκαν βελτιώνουν αυτή την πολύ καλή έκθεση. Θα ήθελα να συγχαρώ και στους συναδέλφους, ε, τους δοσογήτρες. Ε, νομίζω ότι με πολύ καλό τρόπο ε, συντάχθηκε η έκθεση αυτή, γιατί εγώ είμαι εισηγήτρια από την Επιτροπή ΙΦΑΜ και είχα κάποια δυσκολία να παρουσιάσω τροπολογία για τη βελτίωση. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητη αυτή η έκθεση απέναντι στο θέμα της ισότητας των διφύλων. Εγώ προσωπικά έχω παρουσιάσει 12 τροπολογίες και βεβαίως ορισμένες εξ αυτών ήδη αναφέρθηκαν η 86 και 89, η 86 είναι πολύ σημαντική και θα ήθελα η Κομισιόν να βρει την νομική βάση και να τις περιλάβει αυτή στο κείμενο γιατί αναφέρεται στα πλέον ευάλωτα θύματα και φυσικά στην ανάγκη να υπάρξει συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και να αναλυφθούν κατάλληλες δράσεις για να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και επίσης αναφέρεται και στις υποχρεώσεις των κρατών μελών απέναντι στα θέματα που όχι μόνο χρειάζονται προστασία αλλά και βοήθεια και υποστήριξη. Και φυσικά οι ανάγκες των θυμάτων θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο του συστήματος του δικαστικού Σύμματο Δικαιοσύνη, με συγχωρείτε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν εφαρμόζεται ο κανονισμό, τα κράτη-μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα κόμματα και τι ε, αρχέ ε, που αναφέρονται στη Σύμβαση του 89 για την εξάλληψη κάθε είδου διάκριση κατά των γυναικών. Αυτό το έχουμε συμπεριλάβει σε μία από τι τροπολογίε, καθώ ε, και κάποιε άλλε συμβάσει, όπω η Σύμβαση τη Χάγη για την προστασία των παιδιών. Και η τροπολογία 89, εκεί τονίζεται η ανάγκη για συγκρίσιμες στατιστικές δεδομένα για ε, τα θύματα της τρομοκρατίας. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό και αυτή η τροπολογία είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο γιατί αν δεν υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα δεν μπορούμε να έχουμε τις ε, αξιόπιστες, τις κατάλληλες στρατηγικές για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα θυματοποίησης των γυναικών. Και θέλω να επαναλάβω ότι η εκθέση αυτή είναι πάρα πολύ καλή και συγχαίρω τις δύο συγκεκριτές για το έργο τους. Τους δύο συγκεκριτές για το έργο τους. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Λίχτενμπέργκερ. Ευχαριστώ. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συνεργασία μα στην υπόθεση αυτή, η οποία χρειάζεται, έχει ουσιαστική σημασία για την υπόθεση αυτή. Η ερώτησή μου λοιπόν προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η εξή. Ποια δυσκολία επακριβώς διαπιστώνεται ως προς την νομική βάση και θα μπορούσατε ενδεχομένως να δώσετε κάποιες απαντήσεις από πλευράς νομικής επιτροπής για το θέμα αυτό. Ερωτώ λοιπόν ποιο ακριβώς το πρόβλημα και σε ποιο βαθμό είναι ή μη επιλύσιμο. Έχω μια κάποια ιδέα φυσικά, αλλά θα ήθελα να ενημερωθώ επακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χιμένας, παρακαλώ. Θα ήθελα, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τον κύριο Αντώνιο Λόπες Ιστούρης, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να παραστεί σήμερα στη ζήτησή μας, αλλά δούλεψε πάρα πολύ σκληρά για την υπόθεση των θυμάτων αλλά και την επαρβάναβα να ευχαριστήσουμε. Και επίση θα πρέπει να σας πω ότι αυτή η έκθεση είναι πάρα πολύ σημαντική. Τα, ε, το, το, το, το οποίο τώρα ξεκαθαρίζεται όσον αφορά την προστασία των θυμάτων. Και εγώ είχα ασχοληθεί επίση τον ε, Δεκέμβριο με μια έκθεση που αφορούσε τι ποινικέ διαδικασίε. συμφωνήσαμε όσον αφορά τι ε, ε, διαδικασίε αστικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και για το, την ποινική διαδικασία. Και είπαμε τι δέσμετρο θα πρέπει να υπάρχει προς χάρη των θυμάτων. Και γι' αυτό και έχουμε και την ε, οδηγία εξασφάλιση των δικαιωμάτων των θυμάτων. Των θυμάτων από Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε στο ίδιο μήκο κύματο, να συνεργαστούμε ε, και στα πλαίσια του τριμερού διαλόγου που έχουμε με Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να έχουμε εργαστή συνεργασία και έτσι να μπορούμε να προτάξουμε ξεκάθαρα αυτό το οποίο ζητάει το Κοινοβούλιο. Ελπίζω επομένω ότι με αυτή την έκθεση θα ξεκαθαριστούν όλα όσα επιθυμούμε και εμείς και η Επιτροπή το, η νομική γιατί πρόκειται για κοινό αγώνα. Την ίδια δεσμεία τον θέλουμε. Και έτσι να υπάρχει ουσιαστική προστασία των, των θυμάτων και να υπάρξει επίσης και πραγματική αναγνώριση των δικαιωμάτων τους. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Λίχτεμπεργκερ για την Επιτροπή. Η Επιτροπή για την κυρία Λεχτινμπέργκερ. Ευχαριστώ. Πολύ καλή ερώτηση βεβαίως. Όχι τόσο ευχέρέ να σα απαντήσω σε αυτό το επίπεδο. Κάποιες, εξηγήσει Κάποιες ίσως θα μπορούσα να σας δώσω, αλλά όχι πλήρη απάντηση, γιατί δεν έχει καταλήξει και η νομική μας υπηρεσία. Η αρμόδια για τις αστικές υποθέσεις, που όπως φαντάζεστε έχει και πολλή δουλειά αυτόν τον καιρό. Θα πρέπει να τους πιέσω και άλλο μάλλον. Η δυσκολία λοιπόν ως προς την νομική βάση έγκυται στο γεγονός ότι στο πακέτο αυτό συγκρίνουμε αφενός με ένα μέσο, ένα νομοθέτημα αστικού χαρακτήρα, την αμοιβαία δηλαδή αναγνώριση και γνωρίζετε κι εσείς ε, τι χαρακτήρα έχουν συνήθως αυτά τα νομοθετήματα, είναι πολύ τεχνικού χαρακτήρα. Αφετέρου δε υπάρχει μια οδηγία η οποία ομιλεί περί εναρμόνισης των ελάχιστων προδιαγραφών στο ουσιαστικό δίκαιο. Και άρα είναι τελείως διαφορετική νομική προσέγγιση. Τα θύματα προφανώς είναι πάντα στην ίδια κατάσταση και προφανώς και θα πρέπει πάντα να έχουν τα ίδια δικαιώματα. Απανταχού δεν έχει καμιά αμφιβολία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς αυτό, κανέναν ενδιασμό, φαντάζομαι το και τα κράτη-μέλη. Αλλά δεν μπορούμε να βρούμε ενιαία βάση νομική, δεν μπορούμε να εναρμονίσουμε δηλαδή ελάχιστες προδιαγραφές, γιατί δεν υπάρχει νομική βάση για εναρμόνιση στο ουσιαστικό δίκαιο. Ε, θα κοιτάξουμε πάντως το θέμα αυτό με όσο το δυνατόν πιο ανοιχτό πνεύμα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια διασταλτική ερμηνεία της ε, νομικής βάσης. Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη καλύπτεται. Το θέμα είναι πόσο μπορούμε να ε, επεκτείνουμε, να ανοίξουμε το πεδίο δηλαδή της έννοιας πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Όπως είπα, θα έχουμε πάντα ανοιχτό πνεύμα στην εξετάσταση του θέματος αυτού και θα επανέλθουμε με πιο πολλές λεπτομέρειες αν μπορέσουμε. Παρακαλώ, η κυρία Λίχτενμπέργκερ για να επανέλθει. Αν μου επιτρέπετε να επανέλθω, ξέρω ότι ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε διάφορες ένομες τάξεις, το αστικό δίκαιο δηλαδή, ε, είναι αυτό της αμοιβαίας αναγνώρισης που βαίνει με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, γραφειοκρατία ε, και ακριβώς για, την, ε, για το σκοπό της προστασίας των θυμάτων υπάρχει ο κίνδυνος Εάν αυτή η διαδικασία μεταφράσεις, γραφειοκρατία, συνεργασία μεταξύ των αρχών προχωρεί με μεγάλη βραδύτητα και γραφειοκρατία να φτάνει τελικά και με μεγάλη καθυστέρηση και να μην εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο ε, υφίσταται νομίζω ότι θα βοηθούσε πολύ στην έννοια και της ευρωπαϊκής ηθαγένειας, στην οικοδόμηση του αισθήματο της ευρωπαϊκής ηθαγένειας, ιδιαίτερα το θέμα αυτό. Και γνωρίζω ότι υπάρχουν κράτη-μέλη αρκετά στα οποία εκδηλώνονται σημαντικές αντιστάσεις ως προς το τι θα μπορούσε να αποτελέσει ή να εννοηθεί ως επέμβαση στο ιστορικό αστικό δίκαιο. Σε όλους τους τομείς έχουμε δυσκολίες, αλλά στην προστασία των θυμάτων έχει ιδιαίτερα τραγικές συνέπειες αυτό. Διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με τον κίνδυνο για το θύμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί ταχύτητα και που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να ε, περιπλακεί μέσα σε γραφειοκρατικούς δεβάλους. Όπως υπόθηκε λοιπόν, και νωρίτερα. Εμείς το παρακολουθούμε. Η Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων ξέρουμε ότι έχει και πρωτοβουλίες του συναδελφού Μπερντλιγκέρε, παραδείγματι από την Ιταλία και πάνω απ' όλα, με στόχο την ανάπτυξη αισθήματος εμπιστοσύνης μεταξύ των σωμάτων, των θεσμών που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Με μια κοινή κατάρτιση, με ενημέρωση αμοιβαία για τα δικαιϊκά συστήματα, όλα αυτά που αποτελούν προϋποθέσεις για να λειτουργήσει ουσιαστικά στην πράξη δηλαδή το σύστημα αυτό της αμοιβαίας αναγνώρισης. Αλλά πάνω απ' όλα είναι επίγον όπως είπα ε, για την προστασία του θύματος, γιατί υπάρχουν κίνδυνοι, απειλή, ε, πιέζει ο χρόνος πολύ συχνά και γιατί Όπως άλλωστε αναφέρεται και στη τελευταία φράση του κειμένου, ε, έχουμε να, ε, απαιτείται και η ορθή ε, εξέλιξη της διαδικασίας αλλά και η αποτελεσματική προστασία του θύματος. Σε αυτό θα ήθελα να μείνω, να το υπογραμμίσω και να συζητήσουμε, γιατί βέβαια όλοι έχουμε πιστεύω κοινέ προθέσεις και στόχευση, σε ποιο βαθμό μπορούμε να βρούμε συμφωνία και σε επίπεδο Συμβουλίου για την προστασία στην αστική υπόθεση. Προστασία του θύματος δηλαδή ε, σε περίπτωση αστική, σε υπόθεση αστική, να μην θεωρηθεί από το κράτος μέλος ως μία επέμβαση στα εσωτερικό του και στην ένωμή του τάξη. Αλλά ε, να πείσουμε ότι είναι χρήσιμη και ότι μπορεί να εξελιχθεί χωρίς ε, δυσκολίες για να μην έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Αυτή είναι η κυρία μου ανησυχία. Όλοι χρειαζόμαστε. Χρειάζεται να αναλάβουμε τις επαφές με τα κράτη-μέλη, τις αρχές, τις εθνικές του ο καθένας, για να καταστήσουμε σαφές ότι δίνεται κακή εντύπωση εάν για λόγους γραφειοκρατικούς, αν, λόγου, αν για λόγους συστημικής του δικαίου καθυστερεί η παροχή προστασίας σε θύματα ε, στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα κοιτώ να δω αν θέλει κανείς άλλο το λόγο. Όχι από ό,τι βλέπω. όπως και να έχει, βλέπω ότι οι συνάδελφοι μάλλον συμφωνούν ως προς τις τοποθετήσεις. Και έτσι όταν έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και το Συμβούλιο. Ελπίζουμε ότι θα εξελιχθεί καλά και αυτή η συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, μεταξύ μας συμφωνούμε. Αυτό είναι το βασικό και μπορούμε να είμαστε και αισιόδοξοι. Αν μου επιτρέπετε τώρα, θα σας δώσω την ε, ενημέρωση τη σχετική με τη διαδικασία. Έχουμε μια ενδεικτική ε, ψηφοφορία. Αλλά κυρία Παβάνοβα, θέλατε το λόγο, στο συγγνώμη αν σας ξέχασα. Για να δευτερολογήσω, για να καταλήξω κάπου, για να μπορέσω να διαβεβαιώσω όλου του συναδέλφου οι οποίοι τοποθετήθηκαν και είπαν για αυτό το διστάγμο, των κρατών μελών, όπω τα είπε και η Ευρωπαϊκή Τροπή, ότι με αυτή την έκθεση προσπαθούμε να μην υποκύψουν στον πειρασμό του να επιβάλλουμε την επιβολή συνταγής κάποιου κράτους μέλους εις βάρος ή πάνω σε άλλο. Απλώς. Να δώσουμε την ευκαιρία σε κάποιον να προστατευτεί με κάποιο οπλοστάσιο μέτρων που υπάρχουν στο κράτος μέλος το οποίο βρίσκεται αυτό το πρόσωπο, το θύμα. Είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και το πρόσωπο αυτό με τα μέσα προστασίας όσον αφορά... Δεν υπάρχει ενιαία τέλο πάντων κάλυψη, ενιαία ρύθμιση. να μην υπάρχει υπάρχουν διαφορετικέ αντιμετωπίσει όσον αφορά την προστασία, τα δεθμιλή δικαιώματα, ό,τι χρειάζεται το αυτό το πρόσωπο. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε ούτε να επιβάλλουμε κάτι σε κάποιο κράτο μέλο. Εκεί που κάποιο παρίσταται για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα όσον αφορά τα μέτρα προστασία. Ελπίζω ότι αυτό θα διασκεδάσει του φόβου το που θα έχουν ενδεχομένω έχουν τα κράτη-μέλη. Ο πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Η ψηφοφορία προσανατολισμού θα λάβει χώρα στις 30 Μαΐου. Vår processen vidare och eh, därmed så då kan vi även eh, avsluta den här ärendet. Και ο φακελός αυτός θα ακολουθήσει την περαιτέρω πορεία του. Τώρα, η συνεδρίαση των συντονιστών ε, θα ξεκινήσει στις 6 ακριβώ ε, εδώ στην αίθουσα αυτή. Και το τελευταίο που ήθελα να πω είναι ότι αύριο θα ξεκινήσουμε την ψηφοφορία στις 9 ακριβώς. Ε, δεν θα ξεκινήσουμε 9 και 5, 9 και 10, θα ξεκινήσουμε 9 ακριβώς αύριο το πρωί. Σας ευχαριστώ.